Mes chers collègues. Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε συγκεντρωμένοι όλοι. Ναι. Θα ξεκινήσουμε. Κυρία Κραπίνη, είστε καλά. Ωραία. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Λούντγκρεν ε, σχετικά με την αρχή επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβάτων καθώς επίσης και άδειε οδήγησης. Ε, κύριε Λούντγκρεν, θα σας δώσω τον λόγο, μετά θα δώσω τον λόγο στους Σκιώδης και μετά θα ενοχλήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εκπρόσωπο, ωραία. Και και το καλύτερο το αφήνω για το τέλος. Έχουμε την γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε που είστε και εσείς μαζί μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κύριε Λούντγκρεν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την ε, πρώτη μου έκθεση ε, ίσως και το τελευταίο μου, γιατί έτσι όπως είδαμε να μοιράζονται μεταξύ των δύο πρώτων μεγάλων ομάδων ε, οι εκθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη. Πρόκειται για πρόταση οδηγίας ε, για τις άδειε ε, οδήγησης, καθώς επίσης ε, και την κατάρτιση ορισμένων οδηγών, δηλαδή οδηγών συγκεκριμένων οχημάτων. Ε, ο στόχος της οδηγίας ε, είναι να ε, αυξηθούν τα πρότυπα και οι απαιτήσει όσον αφορά τους νέους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως δε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του κινδύνου από πλευρά των οδηγών έτσι ώστε γενικότερα στους ε, δρόμους να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά όλα αυτά να γίνουν ε, με εντός των ορίων της θεμητή και των απαιτήσεων του θεμητού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προτείνω πολλές αλλαγές, έστω και αν υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Πρώτα απ' όλα, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε ε, σε, στο σύστημα της διαβίου ε, κατάρτισης έτσι όπως έχουμε και στον, στην Σουηδία. Ε, ε, και ε, να υπάρχει παρακολούθηση όσον αφορά όλες τις διαδικασίες κατάρτισης που θα γίνονται από την αρχή μέχρι το τέλος της επαγγελματικής ζωής. Επίσης, θα ήθελα να δώσουμε στα κράτη-μέλη την δυνατότητα ε, να ε, οδηγούνται με ε, δίπλωμα οδήγησης Β τα οχήματα τα οποία έχουν βάρος κάτω από 4.250 κιλά και επίσης και τα ηλεκτρικά. Επίσης, από τη στιγμή που μονάχα στην, ότι έχουμε ιδιαίτερη αύξηση του όγκου του αυτοκινήτου μονάχα λόγω των συσσωρευτών ας πούμε ε, και αυτό ε, για οχήματα μέχρι 150 ε, κιλά. Επίσης να ληφθούν υπόψη ειδικέ ακραίες συνθήκες, βροχή ή υπερβολικό ψύχος κτλ. Εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν σε τέτοιες περιοχές, δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί να βάζουν αλυσίδες. Έχουμε διαπιστώσει ακόμα και στη Σουηδία ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα και πρέπει να το μάθει κανείς ε, πριν ξεκινήσει να οδηγεί στο σχολείο, στην, ε, στην κατάρτιση. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εθνικά ε, μητρώα έτσι ώστε ε, να ε, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των προσόντων του κάθε ατόμου. Επίσης καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται ειδικά παραστατικά και πιστοποιητικά η Κομισιόν, η πρόταση μάλλον της Κομισιόν χρήζει διευκρινήσεων σε ορισμένα σημεία. Ε, ε αυτές ε, οι ασάφειες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες από χώρα σε χώρα. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούντγκρεν Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητάς. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Λούντγκρεν Ως έμπειρος οδηγός έχει αναγνωρίσει την έκθεσή του τις ανάγκες και έχει κάνει και ορισμένες προτάσεις που πραγματικά είναι αναγκαίες. Όπως είπε ο ίδιος ο κ. Σουλονγκρεν, στόχος της οδηγίας είναι να βελτιώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της καταρτήσεως των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, να την κάνει την κατάρτιση αυτή ελκυστικότερη ιδίω για τους νέους και να οδηγήσει σε αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδηγήσεως στις διάφορες χώρες μέλη της Ένωσης. Ως τώρα δεν έχουν διεξαχθεί συνομιλίες στην, ε, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Παρ' όλα αυτά, ήδη από τώρα τάσσομαι θετικά υπέρ της ιδέας οχήματα άνω των 3,5 τόνων να εξαιρούνται από την οδηγία. Με μπαταρίες που θα βοηθήσει να μειωθούν οι εκπομπές του οξυδίων του θερμοκηπίου, ε, αερίων Επίσης σημαντικό θα είναι να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογή οδηγίας αποκλειστούν μάλλον πρόσωπα που ε, περνούν από επαγγελματική κατάρτιση εφόσον πρόκειται για πρακτική άσκηση στις περιπτώσεις όπου συνοδεύονται στο αυτοκίνητο από δάσκαλο οδήγησης ή από αρμόδιο άλλο υπάλληλο της επιχειρήσεως. Ε, νομίζω επίσης πρέπει να τονιστεί περισσότερο η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη και οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες, όχι μόνο για τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και για άλλες χώρες όπου σημειώνονται συχνά χιονοπτώσεις και αυτές συνεπάγονται προβλήματα στην οδική κυκλοφορία. Σχόλια. Η κατάρτιση των οδηγών αυτοκινήτων και χρειάζεται και περαιτέρω κατάρτιση γιατί έχω μιλήσει και με οδηγούς αλλά και με δασκάλους επαγγελματιών οδηγών υπάρχει θεωρία και υπάρχουν και προσφορές ηλεκτρονικά για κατάρτιση που όμως είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να επαληθευτεί εάν ο υποψήφιος πραγματικά μπορεί να κατατιστεί επαρκώς μέσω των ηλεκτρονικών αυτών προσφορών εκπαίδευσης. Και είναι και τα λεγόμενα, οι λεγόμενες ήπιες δεξιότητες, soft skills, πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη. Ε, έχω υπόψη μου ιδίω τους νέους, οι οποίοι χρειάζονται προσόντα τα οποία μπορούν να αποκτήσουν μέσω της κατάρτισης αλλά και της περαιτέρω κατάρτισης. Και οι 35 υποχρεωτικές ώρες ανά πενταετία σε 7 ώρα είναι και αυτή μια απέτηση που προβάλλεται αλλά συχνά πρόκειται την ομάδα των ανθρώπων ηλικίας άνω των 50 ετών. και για ορισμένους από αυτούς θα είναι δύσκολο. Ίσως μπορεί να μειωθεί στο μισό η, η περίοδος αυτή κατάρτισης. και να ε, παραταθεί, να γίνεται σε περισσότερες ημέρες. Υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες τώρα και για γεωργικά οχήματα, για οχήματα που χρησιμοποιούνται στην δασοκομεία. και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Έχω και μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, της Κομισιόν. Εάν δηλαδή δεν θεωρεί ότι θα ήταν δικαιολογημένο, να μην είναι μόνο οι επιχειρήσεις εκείνες που θα αποκλείονται, αλλά και μεταφορές εμπορευμάτων σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Ναι. Επίσης, η προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες, στο νέο περιβάλλον των κατηγοριών Δέλτα, Δέλτα 1, Υπάρχει διαπίστωση ότι η κατηγορία αυτή διπλωμάτων είναι για λεωφορεία άνω των 8 μέτρων μήκους και για λιγότερους από 17 επιβάτες. Όμως μου είπαν ότι σε λεωφορεία μακρύτερα των 8 μέτρων είναι σύνηθες να υπάρχουν 20 θέσεις καθημένων. Ερώτηση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και μήπως προσαρμοστεί ο αριθμός των επιβατών αλλά παραμείνει το μήκος στα 8 μέτρα αλλά να αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών στους 20. Και κατάρτιση τώρα και όταν μιλούμε για εκπαίδευση στην τροχαία κυκλοφορία νομίζω ότι χρειάζεται αντιμετώπιση των προβλημάτων και της αξιολόγησης των κινδύνων στην ε, τροχιά κυκλοφορία, δηλαδή πρέπει να λαμβάνονται αυτά τα πράγματα υπόψη στην εκπαίδευση, αλλά και αντιμετώπιση της επιθετικότητας, για παράδειγμα, αντιμετώπιση του στρες και άλλων παραγόντων που εκνευρίζουν τον οδηγό ή που περισπούν την πρόσοχή του, όπως για παράδειγμα η χρήση κινητών τηλεφώνων. Πράγματα τα οποία συχνά οδηγούν σε πρόκληση τροχιών ατυχημάτων. Το άλλο ερώτημα είναι των αναπηριών που ότι και αυτά εδώ. Εν όλο, πάντως, θεωρώ στο σύνολό, δηλαδή, ότι το έγγραφο του κ. δεν είναι σωστό. Ασφαλώς, στο όνομα της πολιτικής μου, ομάδα, ομάδας θα καταθέσω συγκεκριμένε τροπολογίες. Νομίζω πάντως ότι ε, δεν θα αμφισβητηθεί η ε, έκθεση, διότι όλοι από τη δημαξία στην κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών. Κύριε Γραπίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ αισιόδοξη σχετικά με την πορεία της εκθέσεως για δύο λόγους. Πρώτα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Κομισιόν έχει προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας από το 2003 και έχει αναγνωρίσει ότι επισημαίνονται ορισμένα προβλήματα. Καλό είναι που προσπαθούμε να τα διευκρινίσουμε τα πράγματα αυτά. Αφενός έχουμε μια ανασφάλεια, μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου λόγω των διαφόρων εξαιρέσεων. Υπάρχουν δυσκολίες οι οδηγοί να επιτύχουν αναγνώριση των ε, προσόντων τους, των τυπικών προσόντων τους. Επίσης υπάρχουν και προβλήματα σχετιζόμενα με την ηλικία. Η συνάδελφός μας του Λαϊκού Κόμματος σωστά είπε ότι ο κ. Λούντκρεν είναι ειδικό άνθρωπος του τομέα αυτό. Και πάντως, σίγουρα, στις συναντήσεις μας με τους άλλους και οδησηγητές, θα υπάρχει κίνδυνος άνθρωπος που προέρχεται από τον χώρο να είναι κάπως υποκειμενικός και να προσπαθήσει να σπρώξει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που ίσως να προκαλέσει δυσκολίες. Εγώ έχω ερώτηση προς την Επιτροπή, την Κομισιόν δηλαδή, και προς τον εισηγητή. Προς την Κομισιόν. Θεωρείτε ότι χρειάζεται διευκρίνηση της μη εμπορικής, ε, των μη εμπορικών μεταφορών. Δηλαδή υπάρχουν περιστάσεις όπου μια χώρα, σε μια χώρα μέλος μάλλον ένα είδος μεταφορών θεωρείται δεν είναι εμπορικές μεταφορές ενώ άλλη χώρα μέλος τις θεωρεί ότι είναι εμπορικές μεταφορές. Εδώ λοιπόν ανοίγεται μια ευκαιρία για να διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά τον κώδικα 95. Ορισμένες χώρες μέλη εγγράφουν τον κώδικα 95 στις άδειε οδηγήσεως. Άλλες τα γράφουν στο πιστοποιητικό προσόντων. Άλλες τα γράφουν αλλού. Νομίζω ότι χρειάζεται μια συνεκτική θέση όσον αφορά αυτόν τον χαρακτηρισμό κώδικα 95. Η έκθεση δείχνει ότι χρειάζεται και μια ε, ε, ενιαία προσέγγιση στα ε, τυπικά προσόντα. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον εισηγητή. Προσωπικά ποτέ δεν κατάλαβα τις τροπολογίες υπαριθμών 3 και 4 που αφορούν το πεδίο εφαρμογή. Και επίσης στην τροπολογία 12 ο εισηγητής ζητεί να εισαχθεί νέου είδους εξαίρεση. Αφενός δηλαδή ο εισηγητής θέλει να αρθεί μια εξαίρεση αλλά στην 12 θέλει να εισαγάγει νέα εξαίρεση. Ίσως τώρα να μην είναι σωστός χρόνος για να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχει ακόμα κατανοήσει πλήρως η πολιτική μου ομάδα. Πάντως ελπίζουμε ότι με την έκθεση του κ. Λούντκρεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση των απαιτήσεων για ε, την κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ε, να ξεκαθαρίσουμε τους ορισμούς και αυτά που είπα προηγουμένω για μη εμπορικέ μεταφορέ. Πρέπει να μιλήσουμε και για τα 4.250 κιλά, 4,25 τόνου, για να αυξήσουμε την ασφάλεια στι εμπορικέ μεταφορέ. Θα επανέλθω και με άλλε λεπτομέρειε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένω και ο εισηγητή μα, αν έχει να προσθέσει κάποια πράγματα, διότι εγώ εμπιστεύομαι τη γνώμη του, αφού είναι και εμπειρογνώμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Λουντκριν για αυτή την ε, πρόταση. Η δική μου η πολιτική ομάδα ακολουθεί την προτινόμενη τροποποίηση. Πρέπει να συζητηθούν οι εξαιρέσει όσον αφορά την περαιτέρω εκπαίδευση και τα θέματα ασφάλειας και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Επίσης έχουμε και να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν όσον αφορά τα ψηφιακά εργαλεία και την ηλεκτρονική μάθηση. Πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά. Η ηλεκτρονική μάθηση οδηγεί σε πάρα πολλές ερωτήσεις κατά πόσον ε, πράγματι μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες ή όχι. Κυρίως αν η ηλεκτρονική ε, κατάρτιση είναι υποχρεωτική γιατί αυτού του είδους η κατάρτιση δεν ολοκληρώνεται με εξετάσεις. Άρα δηλαδή δεν μπορούν να πιστοποιηθούν οι γνώσεις και ε, δεν μπορεί να πιστοποιήσει κανείς ότι ο ε, καταρτιζόμενος έχει οικειοποιηθεί και εφομοιώσει τις γνώσεις. Ε, ο στόχος των προτάσεων είναι βεβαίως η ελαχιστοποίηση του κόστους και η απλούστευση της πρόσβασης στην κατάρτιση. Όμως ε, οφείλουμε να δούμε και την συμπεριφορά των οδηγών στην πραγματική οδήγηση. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι χρήσιμη αυτή η κατάρτιση. Κατά δεύτερον, η ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας. Αυτή η οδηγία προβλέπει ότι οι εθνικές ε, ρυθμιστικές ε, αρχές οφείλουν να ε, εκδίδουν ένα πιστοποιητικό για τους οδηγούς, αλλά σε πολλά κράτη δεν ισχύει αυτό. Για μας το καλύτερο από όλα είναι αντί για 18 μήνες να μιλάμε για 24 μήνες. Και ελπίζω ε, να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική, συμβιβαστική πρόταση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιλμπάου. Eh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η αξιολόγησή μας ε, της, ε, όσον αφορά την ε, τροποποίηση των δύο κειμένων του 2012-2016, η γενική αξιολόγηση, λέω, είναι θετική. Πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίε οδηγοί όντω θα πρέπει να κατακτίζονται σωστά και αυτό είναι ένα στόχο τον οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Συμφωνούμε επίση με την πρόταση εκεί που λέει ότι θα πρέπει να ε, στην ε, διαρκή εκπαίδευση να υπάρξει και η διάσταση της οδικής ε, ασφάλειας γιατί είναι θέμα το οποίο ήδη έχουμε συμπεριλάβει και σε άλλα κείμενά μας που αφορούν και τα σχολεία και τα λοιπά. Επίσης αυτή η κατάρτιση θα πρέπει να είναι όσο γίνεται ε, πιο ε, κατάλληλη για το είδος της δραστηριότητας ε, στο οποίο επιδίδεται ο εργαζόμενος. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ζωτική σημασίας και επίσης θα πρέπει με την χρήση νέων τεχνολογιών να αποκτήσουμε περισσότερη ευελιξία. Θα πρέπει επίσης να δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι δυνατόν να ε, μην προσαρμοζόμαστε στις ε, σπουδές μας, στην εκπαίδευσή μας, στις ε, νέες αυτές τεχνολογίες και να παραμένουμε προσκολλημένοι στο χαρτί και μόνο. Τα ζητήματα τα οποία θίγει ο εισηγητής είναι θετικά, υπάρχει όμως και κάτι άλλο, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει εναρμόνιση όσον αφορά τις ηλικίες γιατί αυτό θα είναι πολύ θετικό. Επίσης ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του, γιατί και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ε, τις τροπολογίες 3 ε, και 4. Εάν ε, η Κομισιόν έχει το έγγραφο, θα ήθελα να έχω την άποψή τους. Αυτά είναι τα ζητήματα επί των οποίων εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας και φυσικά ε, το θέμα και η αναφορά στην αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια δικαίου που πρέπει ε, να υπάρχει σε όλο το τομέα των μεταφορών και ιδίως στους επαγγελματίες οδηγούς. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπάου, επόμενος ομιλητή. Tack ε, Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση είναι ένα κομμάτι της ε, ευρωπαϊκής, της ενωσιακής νομοθεσίας και έχει σχέση με τα φορτηγά. Υπάρχουν βέβαια παραλληλισμοί ε, Έχουμε ε, και την οδηγία για την έκδοση ε, διπλωμάτων οδήγησης ε, και για το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Ο στόχος είναι να αποφεύγονται τα ατυχήματα και να περιστούν κατά το ημίση οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι δεξιότητες των οδηγών, οι οποίες είναι σημαντικές και γι' αυτό λοιπόν είναι εξίσου σημαντικό η οδηγία να προβλέπει τη βελτίωση των δεξιοτήτων των οδηγών. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής. Είναι σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι περτέρω ε, κατάρτιση είναι υποχρεωτική, αλλά ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδίδεται τον τρόπο διήσης φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Και κατά τα άλλα χρειαζόμαστε ε, σαφείς ε, κανόνες για ε, την οδήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύουν σχεδόν παντού τα ίδια κριτήρια. Οι περισσότερες δεξιότητες οδηγούν στην μείωση των ατυχημάτων. Ο κύριος Κράμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ελέγχθησαν πάρα πολλά και κυρίως ε, το ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά πτυχία όσον αφορά τους οδηγούς φορτηγών. Ε, τους οδηγούς των γιοταχή, εκεί τα ρυθμίσαμε τα θέματα, βέβαια τα παλιά ισχύουν όσο υπάρχουν, αυτό κάποιοι το επέκραν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο στο Συμβούλιο. Τώρα όσον αφορά στις εξαιρέσεις, βεβαίως δεν μπορούμε από το 3,5 να πάμε στους 4,3 τρεις και αυτό πρέπει να το αιτιολογήσουμε. Και μόνο για ε, κάποιους συγκεκριμένους τύπους αυτοκινήτων. Ε, η Κομισιόν θα πρέπει να το εξηγήσει, να υπάρχουν εξαιρέσεις, ας πούμε για τα ηλεκτροχήματα, γιατί είναι βαριές οι μπαταρίες. Να υπάρχει κάποια εξήγηση και κάποια εξαίρεση. Και υπάρχει μια επιστολή προς την Κομισιόν το Απριλίο αυτού του έτους και μέχρι τώρα δεν λάβαμε καμία απάντηση. Δεν ξέρω ε, πώς το κατανοεί αυτό η Κομισιόν, αλλά το να μην απαντάς καθόλου αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Ευχαριστώ, κύριε Κράμερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής και της ε, Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής. Κύριε Σίμος, έχετε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά λοιπόν την γνωμοδότηση της Επιτροπής, η γνωμοδότηση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα στις 31 ε, Μαΐου Ε, είναι λοιπόν η άποψη αυτή της Επιτροπής, η οποία δεν μπόρεσε ακόμα να λάβει υπόψη της, ε, τη γνωμοδότηση. Σε μεγάλο βαθμό περισσότεροι συμφωνούν και δεν νομίζω ότι εκπλήσει κανέναν αυτό, διότι η Επιτροπή εκπροσωπεί και την ε, οργανωμένη μεσαία τάξη. Εκπροσωπεί Επιτροπή, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σε εμά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζονται όλες αυτές οι απόψεις όπως και συνδικαλιστικοί φορείς. Ε, εμείς λοιπόν γνωρίζουμε όλα τα πρακτικής φύσεως προβλήματα. Σε γενικές γραμμές εμείς στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής, είναι ισορροπημένη. Πράγματι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα στεγανό σύστημα για να έχουμε πτυχία που δεν είναι παραποιημένα και όλα αυτά τα χρειαζόμαστε έτσι ώστε το σύστημα να είναι αξιόπιστο. Έχει κατατεθεί και η πρόταση, το λέει αυτό και ο συγητής, να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων. Συμφωνούμε εμείς με την πρόταση αυτή και πέρα από αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και ευελιξία. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα, παρακαλώ πολύ να το προσέξετε. Το θέμα αυτό αφορά τον αριθμό των εξαιρέσεων. Δηλαδή, ε, αν έχει ακολουθήσει κανείς ε, έναν, ε, ένα κύκλο μαθημάτων που ασχολείται με την επισήμανση των κινδύνων, η Κομισιόν αποφάσισε σε αυτή την περίπτωση να μην προβλέπονται εξαιρέσεις. Αλλά εγώ αυτό το θεωρώ επικίνδυνο και θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το Κοινοβούλιο να με έτσι ώστε και στον τριμερή διάλογο να υπάρχει και γι' αυτό εξαίρεση. Ως καθηγητής πανεπιστημίου εγώ θα ζητήσω εξαίρεση, μάλλον θα αρνηθώ θα ζητήσω εξαίρεση για έναν φοιτητή που έχει ε, επισκεφτεί κάποιο άλλο πανεπιστήμιο και μπορεί να το πιστοποιήσει. Απευθύνομαι στον εισηγητή και στους ε, οι εισηγητές. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία λείπουν. Υπάρχουν τέσσερα σημεία ε, τα οποία εξετάστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για το 3-1 της ε, γνωμοδότησής μας για τις ε, βασικές δεξιότητες. Πρόκειται καταρχήν για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή ισχύει το εξής. Το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα ε, στο κύκλο μαθημάτων ή ε, μικρές ή μεγάλες εξετάσεις. Εμείς προτείνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιούν και τις δύο αυτές δυνατότητες. Νομίζω αυτό είναι πολύ εύκολο να ρυθμιστεί. Υπάρχει και μία τροπολογία για τις άδειε οδήγηση και για τις ηλικιακές ομάδες. Το και πρέπει να μετατραπεί σε ή διαζευκτικό ή και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Ε, τα ε, άλλα τρία θέματα αφορούν την ε, δομή της εκπαίδευσης στο σημείο 4-7 πρόκειται για τα, τις 7 ώρες μαθημάτων, ολοήμερα μαθήματα για να συμπληρωθούν οι 35 ώρες και αυτά τα ολοήμερα μαθήματα ε, εκεί θα πρέπει να δείξουμε κάποια ευελιξία μπορούμε να τα μοιράζουμε και σε δύο ημέρες ακόμα και ένας φοιτητής πανεπιστημίου ε, το κατά το μέγιστο που μπορεί να συγκεντρωθεί είναι 20 λεπτά. Δεν πρέπει λοιπόν να υπερβάλλουμε όσον αφορά τη διάρκεια των μαθημάτων ε, και κυρίως εφόσον μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι και εξοικειωμένοι με μαθήματα. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε την ευελιξία. Όσον αφορά τώρα την ηλεκτρονική κατάρτιση. Νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε ήδη. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφήνεια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην προβαίνουν σε διαφορετικές ερμηνείες. Ε, θα πρέπει για την ηλεκτρονική κατάρτιση να ορίζεται επακριβώς και ο αριθμός των απαραίτητων ορών κατάρτισης. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια ε, στις μεταφορές, εδώ ο ορισμός πρέπει να είναι εκτενέστερος Δηλαδή, μία ολόκληρη ημέρα να γίνονται μαθήματα όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά και για την υγεία και για την ε, ορθολογική χρήση των καυσίμων. Πολύ ωραία, κύριε Σίμων, σε αυτά που μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα άλλωστε και τώρα θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στην κυρία... Στην κυρία Γιαννίδου. Πολύ ωραίο το όνομά σας, πολύ μελωδικό. Ιωαννίδου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Γνωρίζετε ότι από τη δική μας πλευρά η πρότασή μας ήταν πολύ εστιασμένη. Προσπαθήσαμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα σημεία δηλαδή τα οποία δεν λειτουργούσαν καλά στην προηγούμενη οδηγία, δηλαδή αμοιβαία αναγνώριση ε, των προσόντων, σαφήνεια, ε, ασφάλεια δικαίου και ευθυγράμμιση. Ε, πρόκειται για μια απόλυτα εστιασμένη λοιπόν στα στοιχεία αυτά πρόταση. Γνωρίζετε επίσης ότι έχουμε ήδη στο Συμβούλιο επιτύχει συμβιβασμό. Χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι η έκθεση είναι αρκετά ευθυγραμμισμένη με τα όσα έχουμε ήδη επιτύχει σε επίπεδο ε, Συμβουλίου. Μας αρέσει ε, η τροχιά που έχει ακολουθήσει η έκθεση και βεβαίως μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε βελτίωση που προέρχεται από τη δική σας πλευρά και πηγαίνει προς την ε, κατεύθυνση της ε, βελτίωσης, της κατάρτισης, του περιεχομένου της επιμόρφωσης. Ας πούμε, χαιρόμαστε, μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία που αναφέρεται σε ακραία και ευερικά φαινόμενα. Το βλέπουμε πολύ θετικά, αλλά βεβαίως Βεβαίως είμαστε και σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα είχε σαν στόχο την διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, με τρόπο ε, ικανοποιητικό προς τον λόγο κόστους ωφέλους. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά δύο τροπολογίες σας. Ε, εκεί θα θέλαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Πρώτον, η τροπολογία που αφορά την δυνατότητα οδήγησης καθαρών ε, ε, καθαρών οχημάτων με δίπλωμα τάξεως Β και μέχρι ε, βάρος 4.250 4.250 κιλά. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό ε, δεν θα πρέπει να γίνει στην ε, αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Κατά τη δική μας άποψη δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να κάνουμε αυτή την, αγορά, την αλλαγή, γιατί έχουμε ήδη ένα σύστημα εξαιρέσεων το οποίο λειτουργεί καλά ε, έχουμε λοιπόν εξαιρέσει από ορισμένα κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να ε, ε τσεκάρουμε λίγο το σύστημα αυτό πριν αναθεωρήσουμε ε, την οδηγία για την, για την άδεια οδήγηση. Ζητώ συγγνώμη για την επιστολή σας γιατί δεν ξέρουμε που κατέληξε αυτή η επιστολή που στείλατε με τις εξαιρέσεις. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή έτσι ώστε να σας δώσουμε και επιπλέον διευκρινήσεις. Δεύτερη παρατήρηση η πρόταση διασύνδεσης των καταχωρήσεων CPC ε, και να υπάρχει ένα σύστημα σε, πραγματική, σε πραγματικό χρόνο. Βεβαίως, ε, καταρχήν, είμαστε υπέρ. Ε, είναι άλλωστε μία από τις, μία από τις δυνατότητες τις οποίες αξιολογήσαμε στην μελέτη επιπτώσεων. Καταλήξαμε ότι αφενός πρόκειται για μάλλον ακριβή λύση ε, και γι' αυτό δεν την υιοθετήσαμε. Η ιδέα είναι σωστή, είναι καλή, αλλά θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά ε, τον, το τι σημαίνει ε, όλο αυτό το σύστημα σε πραγματικό χρόνο, γιατί είναι ακριβό και θα είναι ακριβό σύστημα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις, αυτές τουλάχιστον που εγώ έχω ήδη καταγράψει και σημειώσει. Είχαμε Μία πρώτη ερώτηση όσον αφορά τις γεωργικές εξαιρέσεις. Όντως, στην πρόταση της Κομισιόν η αρχική ιδέα ήταν μια και στην οδηγία χρόνου ανάπαυσης και, ε, οδη... οδήγησης ε, από τη στιγμή που υπήρχαν εξαιρέσεις για αυτού του είδους ε, τα μηχανήματα θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να ευθυγραμμιστούμε και εδώ γιατί εάν ας πούμε υπάρχει κάποιος ο οποίος οδηγεί 50 χιλιόμετρα ας πούμε για να πάει να πουλήσει στην αγορά τα προϊόντα του και τα φρούτα του θα ήταν λίγο δυσανάλογο το να του ζητούμε να συμμορφωθεί διαμορφωθεί με χρόνους ε, ξεκούρασης κλπ. Ε, τώρα δεν είναι υποχρεωτική η διατύπωση αυτή. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα ε, να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς ας πούμε για τα 50 χιλιόμετρα ε, αλλά όλα αυτά θα γίνονται σε ε, εθελοντική βάση. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά και αν πραγματικά πρόκειται για πρόταση όσον αφορά την ταξινόμηση ανάλογα με το μήκος και τον αριθμό θέσεων. Αυτό δεν ρυθμίζεται πάντως σε αυτό το κείμενο. Υπάρχει μια άλλη οδηγία η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό, επομένως για την ώρα θα το αφήσουμε. Υπάρχει επίσης και ένα ερώτημα σχετικά με μεταφορές μη εμπορικού χαρακτήρα. Προσπαθούμε να το, να το διευκρινίσουμε αυτό. Αναρωτηθήκαμε και εμείς για αυτό το θέμα, αλλά εν τέλει θεωρήσαμε ότι υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου ε, η οποία δίνει ε, συγκεκριμένο ορισμό ε, για τις μη εμπορικές διαδικασίες και αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογίες 3 και 4. Η τροπολογία 3 καλύπτει ε, την ε, μία από τη σύσταση του εισηγητού, ε, δηλαδή την εκμάθηση βάση εμπειρίας και στο χώρο της εργασίας θεωρούμε ότι αυτή είναι μια καλή προσέγγιση της ε, ε, κατάρτισης και ακολουθεί μάλιστα και το, το παράδειγμα της ε, Σουηδίας κανένα πρόβλημα και η άλλη τροπολογία για τα γεωργικά οχήματα τα καλύψαμε και αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα εσείς και Λούντγκρεν θα σας δώσω το λόγο αλλά πρώτα έχω μια μικρή ερώτηση. Για την άδεια οδηγήσεως για παράδειγμα, ένας μεταφορέας. Μια στιγμή. Ο κ. Λοτοσχίχ μίλησε πριν, είπε πριν, ότι υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα για την αδειοδίκηση. Ως ένας μεταφορέας με βαθμούς, ε, ακόμα και αν χάσει βαθμούς του μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί. Τι γίνεται εκεί. Κανονικά θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Σας δίνω ξανά το λόγο κύριε Lundgren. Από όσο γνωρίζω, όχι. Απαντώ αρνητικά στην ερώτησή σας. Όχι λοιπόν, δεν θα μπορεί να οδηγεί. Να έρθω λίγο στις μη εμπορικές μεταφορές. Το πρόβλημα είναι, στην Σουηδία έχουμε ένα ιδιαίτερο σύστημα για τις μεταφορές. Έχοντας οι οδηγοί μάθει τα βασικά για την οδήγηση του φορτηγού μετά πρέπει να μάθουν την καθημερινή δουλειά. Και γι' αυτό χρειάζεται να συνοδεύονται από έμπειρο οδηγό. Αυτό γίνεται βέβαια στις εμπορικές εταιρείε μεταφορών. Εάν παραμείνουμε τώρα πολύ αυστηροί με τις μη εμπορικές μεταφορές, αυτό σημαίνει ότι καταργούμε αυτή τη δυνατότητα για τους νέους και τις νέες που εκπαιδεύονται ως οδηγοί δεν θα μπορούν να έχουν αυτή την εμπειρία. Και εδώ μιλούμε για 600 ώρες, μέχρι 600 ώρες που μπορούν να μαθαίνουν να οδηγούν με τη συνοδεία έμπειρου οδηγού. Δεν παίρνουν τη δουλειά του άλλου οδηγού. Ο άλλος οδηγός κάθεται δίπλα τους, πληρώνεται και λίγο παραπάνω για να παίξει το ρόλο του εκπαιδευτού και κρατεί και ημερολόγιο για την εξέλιξη του εκπαιδευομένου. Καθημερινού, καθημερινές δεξιότητες του οδηγού του φορτηγού αυτοκινητού είναι πολύ σημαντικές, διότι κάθε μέρα έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικά φορτία, με διαφορετικό βάρος, με διαφορετικό σχήμα. Είναι πολύ σημαντικό. Αν το διακόψουμε το σύστημα αυτό, σημαίνει τότε ότι οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να πληρώνουν για να αποκτήσουν την εμπειρία αυτή. Και ήδη η άδεια οδηγήσεως φορτηγού είναι πανάκριβη σήμερα. Θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώσουν για μερικέ εκατοντάδε ώρε διδασκαλία θα είναι απολύτως δυνατόν πλέον να βρεθούν νέοι οδηγοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. σε ό,τι αφορά την αύξηση της μάζας του φορτηγού από τα 3,5 τόνους σε 4,25. Μιλούμε εδώ για την προσθήκη των συσσωρευτών, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να βρούμε τρόπους διανομής των αγαθών, των εμπορευμάτων δηλαδή, μέσα στα αστικά κέντρα και εκεί το ηλεκτρικό ε, φορτηγό αυτοκίνητο είναι το καλύτερο. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι πολλοί από τους οδηγούς αυτούς έχουν μονάχα άδεια οδηγήσεως τύπου Β, που σημαίνει ότι μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητα, φορτηγά αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνων μεικτού βάρους. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις ε, ε, επιχειρήσεις μεταφορών να βρουν οδηγούς κατηγορίας Γ σε για να μπορούν να οδηγήσουν βαρύτερα οχήματα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και περισσότερο από αυτό. Πιστεύω όμως ότι επειδή η περιβαλλοντική διάσταση είναι πολύ σημαντική σήμερα, νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε την αύξηση της συνολικής μάζας του φορτηγού σε 4.250 κιλά, με εξαίρεση βέβαια μόνο για τα ηλεκτρικά ε, φορτηγά οχήματα. eco-driving, ε, τρόπος δηλαδή περιβαλλοντικός, ε, ε, ε περιβαλλοντικής και ε, συλλογή εμπειρίας κλπ. Και ως πρώην επαγγελματίας οδηγός οφείλω να πω ότι ήταν σημαντικό το μέρος αυτό, αλλά δεν είχα απολύτως καμία ε, χρησιμότητα από αυτό. Για όλα τα υπόλοιπα τα γνώριζα. Αλλά εξεπλάγει όταν έκανα το πρώτο test drive με τον εκπαιδευτή ε, δίπλα μου, και οδήγησα το φορτηγό αυτοκίνητο όπως οδηγούσα κανονικά. Και μετά με έβαλε να κάνω καινούριο test drive με τα σχόλια του εκπαιδευτού μου. Έλεγε τώρα κάνει αυτό, τώρα κάνει εκείνο. Και εξεπλάγει πραγματικά πόσο εύκολο ήταν να μειώσει κανείς την κατανάλωση καυσίμου με μικρές αλλαγές της οδηγικής μου συμπεριφοράς. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και τουλάχιστον στη Σουηδία αυτό εντάσσεται στην περιοδική κατάρτιση των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων. Θα κάνουμε συναντήσεις βέβαια με τους σκιωδησηγητές και η ελπίδα μου είναι η πρώτη συνάντηση των, των σκιωδών να γίνει πριν από τις θερινές διακοπές και να επανέλθουμε, θα επανέλθουμε για να σου πούμε τις ημερομηνίε. Ευχαριστώ ήδη για τα σχόλια που μου έγιναν και ευχαρίστω να συναντήσω ξανά τους σκιώδεις ηγητές και συγκητές και από όσα ακούω μου φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πολύ θετική συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λοντκρέν για την παρουσίαση τη εκθέσεώ σα, που πραγματικά ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο τον κόσμο και λόγω βεβαίως της επαγγελματική σας ε, καταρτήσεω και λόγω της ε, εθνικότητά σα μα δώσετε καλά παραδείγματα πρακτικών που μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λοντκρέν. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών Λίγη στις 27 έκτου στις 2 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε. με την έκθεση για τις διαμεθοριακές παραδόσεις δεμάτων με συγκίτρια την κυρία Άντερσον και μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδες οδησηγητές καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που έχω τη δυνατότητα να, βοηθεί, να ε, συμβάλλω στις ε, των ε, τροπολογιών που έχουμε πολλές, είναι 424 μαζί με τις δικές μου, πολλές είναι πολύ χρήσιμες. Όλοι δηλαδή έχουν εξετάσει την εκθεσή μου έχουν και τεχνικές λεπτομέρειες και για τα, παράρτημα, τα παραρτήματα μάλλον και την καλύτερη σύνταξή τους. Υπενθυμίζω σε όλους και όλους ότι ο κανονισμός αναφέρεται μονάχα σε παραδόσεις δεμάτων διαμεθοριακά. Έχει επομένω σχέση με την ενιαία αγορά, αλλά παρόλα αυτά είναι σωστό η Επιτροπή Μεταφορών να εγκύψει στο θέμα, διότι εδώ υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις για όλο τον τομέα των μεταφορών και logistics και είναι και μεγάλη προτεραιότητα και για μας. Όσον αφορά τώρα τις διαμεθοριακές ε, παραδόσεις δεμάτων και την πρόπτικη, ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες διαμεθοριακής παραδόσεως δεμάτων, διότι πράγματι ακούμε συχνά από καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις ότι δεν απολαμβάνουν καλές υπηρεσίες ούτε και οι τιμές είναι χαμηλές. Όταν ε, παραγγέλουν ή όταν παραλαμβάνουν ε, δέματα. Όμως μόνο, ξαναλέω, για τον τομέα των, της παραδόσεως ε, δεμάτων διαμεθοριακώς. Και βεβαίως υπάρχει εδώ και η οδηγία των καθολικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει στη μελέτη τύπου ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Το ερώτημα, όπω πάντα, είναι πώ θα αντιμετωπιστούν καλύτερα τα προβλήματα αυτά. Δέχομαι ότι δεν θα συμφωνήσουν όλε και όλοι στους τρόπου που προτείνω, αλλά εξετάζω όλε τι τροπολογίε, έχω και έναν αριθμό συμβαστικών τροπολογιών που επεξεργάζομαι και νομίζω ότι όλε και όλοι κάνουμε κάποια πρόοδο. Όσον αφορά ορισμένα από τα θέματα τώρα που έχουν ανακύψει, το βασικότερο είναι το ερώτημα εάν οι κανονισμοί που καλύπτουν, τόσο οι διατάξεις που καλύπτουν τη διαφάνεια των τιμών και την αξιολόγηση των τιμών θα πρέπει να είναι για παρόχους καθολικής υπηρεσίας ή αν θα πρέπει να είναι για να ισχύουν για όλους τους παρόχους παραδόσεων δεμάτων. πάντοτε με την έννοια της διαμεθοριακής πάρδοσης, όπως εξήγησα. Θα χρειαστεί να διεξαγάγουμε κάποιες σοβαρές συζητήσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα. Πάντως είμαι απολύτως και ενθουσιοδός, και υπέρ της εξέβρεσης μιας λύσης που να επιτρέπει ωστόσο και διαφάνεια για την αγορά. Οι ρυθμιστέ διαθέτουν κάποιε πληροφορίε, όμω όχι όλε όσε χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά του και χαίρομαι που πολλέ από τι τροπολογίε το τονίζουν αυτό. Προβλέπουν επίση και προστασίε και λέει ότι οι αξιολογήσει δεν θα πρέπει να είναι σχετικέ με ρύθμιση τιμών, αλλά θα πρέπει να είναι μια πραγματική δοκιμασία και μόνο εφόσον είναι αναγκαίο θα πρέπει να δοθούν και άλλες πληροφορίες για την αγορά παραδόσεως δεμάτων. Το βασικό αυτό είναι το 3 για την παροχή πληροφοριών που εφαρμόζεται, επιβάλλεται τέλο πάντων σε όλους τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και το επίπεδο της πληροφορίας που πρέπει να δίνεται για το συνολικό αριθμό δεμάτων. Κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα απασχολούμενα πρόσωπα, γιατί αλλιώ πώ θα μπορέσει να αξιολογήσει κανεί εάν η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό τη διότι είναι ε, σημαντικό το, ε, ε αυτή τη πληροφορία. Βασικά θέματα που αφορούν τους υπεργολάβους, αν είναι αναγκαίο ή πάντως ενδιαφέρον να δίνονται πληροφορίες και για τους υπεργολάβους και γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους παρόχους χρησιμοποιούν και οι άτομα που εργάζονται υπεργολαβικά και πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται στον τομέα αυτό. Και το άρθρο 3 περιλαμβάνει αυτά τα θέματα στα οποία άλλωστε κατευθύνονται και οι τροπολογίες. Και είναι χρήσιμε οι εισρωέ αυτέ για του συμβάσιμου. Σημαντικό είναι επίση αν θα πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι, ώστε κανένα πάροχος των σχετικών υπηρεσιών να μην είναι να παρέχει πληροφορίες αυτές εφόσον απασχολεί λιγότερο από έναν αριθμό ατόμων και πώς υπολογίζεται αυτό. Ορισμένα από τα πράγματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα, ορισμένα μπορούν να επιληθούν με αρχέ τη απλή κοινή λογική. Ε, με, αυτά θα δούμε στις, συμβαστικέ συμβαστικές τροπολογίες. Θα γνωρίζετε και για τα όρια. Έχουμε όριο, προτινόμενο όριο 10 πρόσωπα, 25 40 και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την δομή των ε, σχετικών επιχειρήσεων των εταιριών. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των τιμολογίων και την αξιολόγηση των τιμολογίων, πάλι εδώ προβάλλονται διάφορες ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να αποδώσει αυτό. Υπάρχει το άρθρο 4, το οποίο προβλέπει ένα δημόσιο τιμολόγιο. Θα πρέπει να ισχύει αυτό για όλους τους παρόχους. Και πάλι, σε ό,τι αφορά την δημοσίευση πληροφοριών, είναι σημαντικό για τους ρυθμιστές να γνωρίζουν εάν οι ιδιώτες πάροχοι παρέχουν και αυτοί οι πληροφορίες για το τι τιμές επιβάλλουν για συγκεκριμένες ε, περιοχές και συγκεκριμένα είδη δεμάτων κλπ. και θα πρέπει να εξετάζονται κάποια συγκεκριμένες, κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δεμάτων, ώστε να είναι πιο δυνατόν να αντιμετωπιστεί από την πλευρά του κανονισμού. Και μιλούμε εδώ για μεμονωμένα δέματα. Δεν είναι λοιπόν bulk tariffs, δεν είναι ε, τιμολόγια που να ισχύουν για μεγάλους όγκους δεμάτων. Ακόμα μένουν πολλά να συζητηθούν. Πάντως το άρθρο 4 πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το 5 και εδώ Πολλοί λένε ότι το 5 πρέπει να καταργηθεί απολύτως. Και ίσως να εφαρμόζεται μονάχα στους παρόχους καθολικών υπηρεσιών. Εγώ είπα ότι αυτό δεν είναι αναγκαία δίκαιο να διαμορφωθεί έτσι ο κανονισμός και μία από τις αρχικές κριτικές απέναντι στην πρωτοβουλία αυτή ήταν ότι στόχευε αυτούς τους παρόχους και δεν λάμβανε υπόψη το ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη δουλειά να κάνουν. Ναι, πράγματι έχουν κάποια δουλειά να κάνουν, αλλά αυτό είναι ζήτημα που εντάσσεται στη συνολική συζήτηση τη ολοκλήρωση τη ενιαίας αγορά, μια έντιμη ενιαίας δίκαιη ενιαίας αγορά που θα προσελκύσει και περισσότερου να συμμετάσχουν στην παροχή υπηρεσιών παραδόσεων δεμάτων διαμεθοριακά, είτε πρόκειται για χρήστε είτε πρόκειται για παρόχου. Πάλι συζητούμε λοιπόν το άρθρο 5 και αν θα πρέπει να παραμείνει και με ποια μορφή πώς μπορεί να βελτιωθεί, πως ενδεχομένως εφόσον δίνονται κάποιες πληροφορίες, τονίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ποιου είδους υπηρεσίες επιβάλλεται, ώστε να απηχείται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχουμε να προστατεύσουμε την καθολική υπηρεσία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιτευχθεί αυτό και με διευκρινήσει που θα γίνουν και στην αιτιολογική, και στην αιτιολογική έκθεση. Υπάρχει λοιπόν αρκετή δουλειά να γίνει ακόμη. Υπάρχει και ένα νέο άρθρο 6 που ορισμένοι 6 μόνο, ξαναλέω, το νέο άρθρο 6, όχι το παλαιό, το οποίο προβλέπει έξτρα προστασία υπέρ των καταναλωτών. Και παρακαλώ όλους να το εξετάσουν. Ορισμένοι το έχουν δει και έχουν υποβάλει και τροπολογίες για την προστασία των καταναλωτών. Προσπαθούμε στην πραγματικότητα να προβλέψουμε μέσα στο νέο άρθρο 6 ιδιαίτερε προστασίε των καταναλωτών και θέματα ποιότητα. Το παλαιό 6 επέβαλε υποχρεώσει στου παρόχου καθολικών υπηρεσιών για να ανοίξουν τα δίκτυά του. με τρόπο που εγώ θεώρησα άδικο δεν υπάρχει τρόπος να ανοίξει αυτό με δίκαιο τρόπο. Και ορισμένοι συμφωνούν μαζί μου ότι καλύτερα ήταν να διαγραφεί. Και ορισμένοι το δέχονται και το κάνουν στις τροπολογίες τους. Και τέλος, οι τελικές διαταξίες, για το πώς θα το δούμε αυτό. Αλλά θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να συνδέεται και με την αναθεώρηση της οδηγίας ταχυδρομικών υπηρεσιών για να μην προκαλέσουμε προβλήματα και πάλι λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις αναθεωρήσεως, υπάρχει κάποιο βαθμό συμφωνίας και δυνατότητα συμβασμού για το πώς θα λειτουργήσει. Πρόκειται δηλαδή για ένα κανονισμό που προσθέτει στα ήδη υφιστάμενα. Δεν αφαιρεί από τους παρόχους καθολικών υπηρεσιών υποχρεώσει, ούτε τους επιβαρύνει. Μπορεί τελικώς να μην καταλήξουμε εκεί, αλλά ασφαλώς αξίζει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ, της, αυτού του κανονισμού επικοδομητικά. Και ελπίζω θα ξαναπούμε τον Ιούλιο. Ευχαριστώ κύριε Άντροσον. Κύριε Φέρμπερ, καλώς ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για την παρουσίαση της διαδικασίας. Έχουμε συνδεθεί ήδη δύο φορές και νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει πια σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι από όλες ε, τις καπνοδόχους θα αναδύεται, θα βγαίνει λευκός ε, καπνός. Δεν νομίζω ότι φτάσαμε ακόμα εκεί. Ε, υπάρχουν οι αρχές όμως επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει και μετά δεν είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Πρώτη βασική αρχή. Σε αυτήν την συγκεκριμένη πρόταση, σε αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό, οι ε, καθολικές υπηρεσίες ε, τι ρόλο παίζουν εμείς δημιουργήσαμε την καθολική υπηρεσία στην οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων έτσι ώστε στην οδηγία περί ταχυδρομείων μάλλον, έτσι αν ζει, είτε ζει σε αστική περιοχή είτε στην επαρχία ή και αν είναι και μόνος του κάπου σε ένα βουνό, αυτό το συζητήσαμε γιατί και πριν από 10 χρόνια, να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίε και μάλιστα σε προσιτό κόστος. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπή αποβλέπει σε όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, δεν διασφαλίζονται οι προσιτές τιμές, αλλά ε, είναι πολύ ακριβό το να στείλει κανείς ε, ένα δέμα πέρα από τα σύνορα. Πολύ πιο ακριβό από ότι μέσα στο ίδιο το κράτος. Ε, αυτό όμως δεν μπορούμε να το δεχτούμε και από αυτού συμφωνούμε όλοι. Τείτε λοιπόν το εξής ερώτημα. Τώρα, εάν συμπεριλάβουμε όλους τους φορείς αποστολής ε, δεμάτων, Δείτε το θέμα του, ε, της καθολικής υπηρεσίας. Ο ανταγωνιστής ε, δεν έχει την υποχρέωση παροχής ε, καθολικής υπηρεσίας. Δεν είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες ε, σε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάποια μειονεκτήματα. Παραδείγματο χάρη δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στο ΕΛΚ ανησυχούμε ότι αν αρχίσουμε τώρα ε, σε ένα σημείο να τα από αυτή την έννοια της καθολικής υπηρεσίας, στο τέλος θα καταλήξουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλει και η ίδια η συγγήτρια και που είναι και ένα κομμάτι της πρότασης της Επιτροπής. Δηλαδή θα καταλήξουμε το να ασχοληθούμε με την αποστολή δεμάτων, δεμάτων με την απασχόληση. Εμείς το μόνο μας που θέλουμε είναι να διευκολύνεται ακριβώς αυτή η δασυνοριακή αποστολή έτσι ώστε να μπορούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου να στέλνουν και αυτές τα προϊόντα τους. Γιατί σε τελική ανάλυση όλοι βασίζονται στην καπελική υπηρεσία. Δεν μπορούν να φτιάχνουν, φτιάχνουν ο καθένα μόνος του ένα φορέα για να στέλνει θέματα. Δεν ήταν εξάλλου αυτός ο στόχος. Όσο λοιπόν γυρίζουμε γύρω από το βασικό θέμα, όσο δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το κέριο θέμα, τουλάχιστον για το ΕΛΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Απλά διότι συγκρούνται δύο βασικές έννοιες για τις οποίες έχουμε ήδη συζητήσει ε, με κατά το παρελθόν, εγώ είχα την εντύπωση ότι είχαμε όμως συμφωνήσει. Γιατί η Ολομέλεια είχε αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία να εστιάσουμε την προσοχή μας στις καθολικές υπηρεσίες. Θεωρώ λοιπόν ότι τίθεται ένα θεμελιώδης ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι το εξή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και διαφορετικέ εμπειρίε από διαφορετικά κράτη-μέλη. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου τα πράγματα πάνε πολύ καλά και άλλα που τα πράγματα πάνε σχεδόν καλά και στο ενδιάμεσο υπάρχουν και πολλά άλλα. Ο καθένα λοιπόν ε, έχει τι δικέ του εμπειρίε, κάτι που δεν διευκολύνει την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα. Και εμείς ε, τα αναφέρουμε στην οδηγία μας ε, σχετικά με την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Πρώτον, οι διασυνοριακές αποστολές δεν μπορούν να είναι πολύ περισσότερο ακριβές από ότι οι εσωτερικές αποστολές. Εμείς ως ΕΛΚ λέμε ναι στη διαφάνεια όσον αφορά στους παρόχους καθολικών υπηρεσιών. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην διασυνοριακή αποστολή δεμάτων. Και επ' αυτού υπάρχουν διαφορετικές ε, διαφορετικοί ορισμοί και αυτά πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Και τρίτον, υπάρχουν κρατημέλη όπου η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή ε, δεν εφαρμόζει τις ε, τα απαιτούμενα των, της οδηγίας ε, περί ταχυδρομείων. Γι' αυτό λοιπόν ε, για κάποιον που ενδιαφέρεται είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί στην αγορά. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διοικητούμε κατά πόσον στις νέο συστηνόμενες επιχειρήσεις να προσφέρουμε ειδική προστασία όπως το έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις ή αν θα πρέπει στις επιχειρήσεις ε, που έχουν και ένα μόνο εργαζόμενο και από τον πρώτο εργαζόμενο να τις ε, υπάγουμε στις ρυθμιστικές αρχές. Ε, με τον τρόπο όμως αυτό παρεμποδίζουμε την πρόσβαση στην αγορά, κυρίως για πολλές νέες επιχειρήσεις και γι' αυτό εμείς ως ΕΛΚ δεν το επιθυμούμε. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ένα κατώτατο όριο έτσι ώστε οι νέο συσταθήσεις επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά πριν ε, αρχίσει να ισχύει και για αυτές ε, η νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν λοιπόν όπου διαπιστώνουμε ότι στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας ε, περί ταχυδρομείων υπάρχουν περιπτώσεις όπου ε, κράτη, όπου τα τρία τέταρτα της επικράτειάς τους ε, τα έχουν ορίσει ως περιφέρεια. Και δεν αναφέρομαι σε κράτη με μεγάλη νησιωτική έκταση. Λόγω αυτού λοιπόν έχουν επιδεινωθεί τόσο πολύ οι ταχυδρομικές υπηρεσίες σε μία χώρα και ο εθνικός, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή παράλληλα απαγορεύει το να συσταθούν νέες επιχειρήσεις. Εμείς όμως αυτό ε, θέλουμε να το ε, λύσουμε. Εμείς έχουμε θέματα που είναι καθοριστική σημασία και πρέπει να επιληθούν. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να ελπίζω ότι στο πλαίσιο των περαιτέρω διαπραγματεύσεων η κυρία εισηγήτρια θα προσπαθήσει να ασχοληθεί με όλες τις προτάσεις έτσι ώστε στο τέλος να καταλήξουμε σε κάτι που θα εξυπηρετήσει εξυπηρετεί τον καταναλωτή. Και τελικά ο καταναλωτής ε, δεν νομίζω ότι εξυπηρετείται από κατακλυσμό πληροφοριών. Ο καταναλωτής ε, χρειάζεται ε, βασικές πληροφορίες, αυτό είναι το ένα. Και κατά δεύτερον, αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές για να μπορούν να εξαλείφονται κακοδαιμονίες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε και με ρυθμίσει στην αγορά. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε και το λέω αυτό εμφατικά και κατηγορηματικά. Δεν πρέπει να υπάρχει μια κακώς ενούμενη διαφάνεια των δεδομένων και με τον τρόπο αυτό να ασκήσουμε πίεση στους παρόχους καθολικών υπηρεσιών που θα είναι καθοριστικά εις βάρος τους. Για να μπορεί ένας ανταγωνιστής να επιβιώσει την αγορά ε, πρέπει να είναι πιο ευνοϊκός, αλλιώς δεν θα τα καταφέρει και να είναι πιο ευνοϊκός παρότι καταβάλει και το ΦΠΑ. Όταν όμως το κάνει αυτό ε, δεν υπάρχουν πολλά σημεία για να μπορεί να εξοικονομήσει κόστος και εάν ο πύχης ε, στον οποίο θα πρέπει κανείς να προσαρμόζεται είναι ο φορέας καθολικών υπηρεσιών, με όλα αυτά το μόνο που κάνουμε είναι κοινωνικό dumping, το οποίο εμείς ως ΕΛΚ δεν το επιθυμούμε. Αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, φτιάξαμε και την έννοια του φορέα καθολικών υπηρεσιών. Σας παρουσίασα ένα ολόκληρο σκηνικό. Μέσα από αυτό είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις ε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε δώσει και γραπτά τη θέση μας ε, στην εισηγήτρια. Θα κάνω και εγώ κάποιες προτάσεις για συγκεκριμένα άρθρα με βάση αυτά τα οποία αποφάσισε η Επιτροπή Κοινής Αγοράς. Δεν τα βρίσκω ανόητα αυτά που αποφάσισε, μπορούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και ελπίζω παρόλα αυτά να κατορθώσουμε στις 11 Ιουλίου να ψηφίσουμε. πάντω αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Φερμπέρα. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να, ζητήσω, ε, να ε, να σας πω ότι ο κύριος Κούν δυστυχώς ε, ζητά συγγνώμη δεν μπορεί να είναι εδώ. Ε, όμως, όμως ε, μπορώ να ε, ε, σας πω ότι έχουμε 20 καλεσμένους από το τοπικό κοινοβούλιο της εκλογικής του περιφέρειας, το Μέκλεμπουργκ της Δυτικής Πομερανίας. Ε, αν κατάλαβα καλά, ε, είναι η βόρειο-δυτική περιφέρεια της Γερμανίας κοντά στη Βαλτική θάλασσα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας καλωσορίσατε και ε, πρέπει να σας πω ότι ε, πραγματικά εμείς θέλουμε να βλέπουμε εκπροσώπους τοπικών ε, κοινοβουλίων και χαιρόμαστε όταν ακούτε προσεκτικά τα όσα κάνουμε εμείς εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο κύριος Λοτόφσκι. Madame la Présidente, ja chciałbym się dołączyć do podziękowań θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Άντερσον γιατί δούλεψε με μεγάλο ενδιαφέρον και αν και βλέπουμε στις ε, τροπολογίες κάποιες ε, θετικές εξελίξεις, παρόλα αυτά βλέπουμε να υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Και είναι κρίμα που η συγγήτρια έλαβε μόνο κάποιες από τις ε, τροπολογίες που καταθέσαμε ως ε, πολιτική ομάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το ότι οι εταιρείε που στέλνουν θέματα ε, πρέπει να καταθέτουν κάποιες εκθέσεις, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις και ως εκ τούτου η οδηγία δεν θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Αναφέρομαι κυρίως σε υπεργολάβους. Αν όμως δεν επισημάνουμε ότι εμείς κάνουμε λόγο μόνο για μεγάλους υπεργολάβους, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η οδηγία. Κάποια στοιχεία ε, αναφέρονται εις διπλούν και νομίζω ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά την όλη εικόνα της αγοράς. Οφείλουμε ε, τις ε, υποχρεώσεις ε, των υπεργολάβων να τις καταστήσουμε πραγματικές. Τώρα, όσον αφορά τις εταιρείε που στέλνουν δέματα και έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, η κυρία εισηγήτρια προτείνει 25 άτομα. Αυτό όμως είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν είναι και συμβατό με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει λόγο για 50 άτομα που είναι πολύ πιο λογικό και δεν θα οδηγήσει και σε μεγάλη επιβάρυνση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έγκριση της τροπολογίας 235 δεν πρέπει να ε, παραλείπουμε και την κατάσταση των καταναλωτών. Ε, αυξάνεται, επιδεινώνεται το ε, διοικητικό άκτος και αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερο σε αύξηση του κόστους. Ε, κατανοώ αυτά που λέει η συγγήτρια στο άρθρο υπαριθμών 5, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Εξάλλου είναι απαραίτητο να υπάρχουν και άλλα, ε, άλλες πληροφορίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις και τα καταληκτικά τέλη. Η τροπολογία μας υπαριθμών 288 δυστυχώς δεν ελήφθη υπόψη και αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι λαμβάνεται μόνο υπόψη η τιμή που αναφέρει ο φορέας καθολικής ε, παροχη καθολικης καθολική υπηρεσίας. Οδηγία 97-67. Κατανοούμε βέβαια ότι η συγγήτρια έχει κάνει πάρα πολλά ε, για να καταλήξει συμβαστικέ ε, προτάσει. Ευχαριστώ. τελεινικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και πρώτα θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Να αρχίσω λέγοντας ή μάλλον τονίζοντας ότι Υπάρχει ένα θετικό αίσθημα ότι όλοι έχουμε τον κοινό στόχο, δηλαδή μια λειτουργούσα αγορά μεταφοράς δεμάτων και βεβαίως ορισμένοι έχουν υψηλότερη αναγνώριση της ανάγκης που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι έχουμε και κάποιο, κάποια ιδέα για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί και στο μέλλον η αγορά παραδόσεως δεμάτων. Δεύτερο, όπως ελέγχθη ήδη από ορισμένους προλαλήσαντες συναδέλφους, πρέπει να εξετάσουμε και το σχέδιο νομοθετήματος και από την πλευρά του κανονισμού e-commerce. Υπάρχουν κάποιες ανομαλίες στην αγορά. Κατανοεί κανείς ότι υπάρχει διαφορά τιμών 7 ε, ποσοστιών μονάδων. Δεν θέλω να αναπτύξω ε, την δομή των ε, των τιμών είναι όμως κατανοητό. Ορισμένοι δεν αναγνωρίζουν τις παραδόσεις ως διαμεθοριακές παρόλο που είναι. Ορισμένες όμως διαφορές είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες. Και άρα υπάρχει λόγος να εξετάσουμε ευνοϊκά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένοι εκφράσαμε αμφιβολίες και εγώ και κάποιο δισταγμό να προχωρήσουμε νομοθετικά στο προκείμενο ε, θέμα βεβαίως διδάσκεται κανείς καθώς προχωρεί. Και φαίνεται, πολλοί stakeholders μας λένε ότι αξίζει να γίνει μια προσπάθεια. Το πιο σημαντικό είναι όμως να διατηρήσουμε το πεδίο εφαρμογή και να συμβάλλουμε ώστε να γίνει συμπληρωματικό στην οδηγία ταχυδρομικών υπηρεσιών και να προσπαθήσουμε να επισκευάσουμε ό,τι πρέπει να επισκευαστεί χωρίς να μπούμε σε, μια, σε ένα ατυχές νομοθετικό εγχείρημα που θα οδηγήσει τελικώς σε στρεβλώσεις της αγοράς και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει. Είμαι σχετικά αισιόδοξο. Βέβαια δεν έχουν προχωρήσει ακόμα αρκετά οι συζητήσεις, αλλά είναι και δύσκολο ο φάκελος, έχει πολλές διακλαδώσεις και εκτιμώ την ε, προσπάθεια της εισηγητρίας να λάβει υπόψη και τις απόψεις άλλων και νομίζω ότι όντω ε, προχωρούμε. Σταδιακά και αργά, αλλά να, αρκεί να είναι σωστά. Ένα στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογή ότι σε μία διετία θα διεξαχθεί αναθεώρηση της οδηγίας ταχυδρομικών υπηρεσιών. Και κάτι που απασχολεί εδώ ορισμένους από εμά και το εντάσσω σε αυτή τη διαδικασία περισσότερο, για να μην δημιουργηθεί ένα είδος ευχολογίου από το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα δηλαδή να, να δημιουργηθεί μια νομοθεσία υψηλής ποιότητας που ε, να εξυπηρετεί την λεγόμενη better regulation, έστω και αν αυτό σας ακούγεται κλεισέ. Θα έχω να πω τα εξής. Άρθρο 4, στο οποίο έγινε αναφορά ορισμένες φορές, Υπάρχουν διαφορές. Το ερώτημα είναι εάν όλοι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καλύπτονται ή μόνο οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών. Οφείλω να πω ότι όπως αναπτύσσεται η αγορά και οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών είναι οι μόνοι που εκπροσωπούν την αγορά αυτή και ενδέχεται Όπω να υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Πολλοί επιχειρηματίες όμως αλλάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και θα αλλάξει και επομένως και η αγορά. Κάτι που είναι σημαντικό και εκτιμώ που το λαμβάνει υπόψη η εισηγητία είναι ότι μειώνουμε την αγορά σε single piece tariff, δηλαδή ε, τιμολόγια για μεμονωμένα δέματα. και ηλεκτρονικούς ε, λιανεμπόρους. Δεν μιλούμε για συμβάσεις μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ειδικέ ρυθμίσεις. Μιλούμε μόνο για μεμονωμένες παραδόσεις. Βλέπω ότι σας διασκεδάζει ο κ. Βαντεκάμπ, αλλά προφανώς δεν διασκεδάζεται με αυτά που λέω εγώ. Το βλέπω, ε, το βλέπω καθαρά. Διακόπτη η πρόεδρο Όχι, εγώ δεν ειρωνεύομαι κανέναν ε, που βρίσκεται μέσα στην Επιτροπή. Έχω ακόμα δύο θέματα. Συνεχίζει ο κ. Τέλιτσκα. Θέλω να υποστηρίξω την πρόταση Επιτροπής για να γίνει το affordability test. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό βασίζεται στο κόστος και το είπαν και ορισμένοι αυτό και χαίρομαι που συμφωνούμε και σε αυτό και το κρατήσατε σαφές η συγκεκριά δεν επιδιώκουμε κρυφές ρυθμίσεις τιμών. Και τα external rates. Και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Γνωρίζει και η συγκεκριά ότι προτιμώ μια ρύθμιση σε δύο βήματα για τις τελικές τιμές. Για το άνθρωπο 6 τώρα και τη διαφάνεια, αυτό θα έχει τις πιο ορατές επιπτώσεις στους καταναλωτές, βραχυπρόθεσμα διότι αυτό ζητεί να ανοίξουν τα δίκτυα σε άλλους μεταφορείς δεμάτων και ιδίω σε εκείνους που δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτούν με μεγάλους επιχειρηματίες, μεγάλους operator. Ορισμένοι θα πούν να τα αφήσουμε αυτά στο εμπόδιο, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Το άνθρωπο αυτό δεν αναφέρεται στην αμφισβήτηση των επενδύσεων ή των μεριδιών αγοράς των παρόχων καθολικής υπηρεσίας. Και εκεί θα ήμουν αντίθετο. Αλλά να μοιραστούν το κόστος του δικτύου. Χρειαζόμαστε όμως κάποιες εγγυήσεις. Τελική παρατήρηση, μάλλον δύο τελικές παρατηρήσεις πολύ σύντομες, αφενός. Παρακαλώ, εάν θέλουμε μια στέρεα συμβιβαστική λύση, ας αποφύγουμε να περιλάβουμε στο νομοθέτημα τα διάφορα θέματα που θα ήθελε καθένας για καταναλωτές κτλ. Έχουμε μια νομοθεσία στην οποία μπορούμε να παραπέμπουμε διαρκώ. και τα θέματα των υπεργολάβων που υπέμψαν ορισμένοι συναδελφοί μας. Έχει την στήριξή μας η συγκήτρια και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε κάποιες περιττές δυσκολίες. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία του Ιουλίου. Ευχαριστώ κύριε Τελίτσκα, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το, λόγο στον κύριο Βίμ Κάμπα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ζητώ Συγγνώμη, γιατί όντως αφαιρέθηκα λίγο. Ε, ίσως γιατί είμαι και ανυπόμονος. Ε, γιατί ήδη ε, δεύτερη εβδομάδα παρακολουθώ αυτό το ε, φάκελο, αυτό το θέμα και έχω την εντύπωση ότι προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα και να συμφιλιώσουμε τα ασυμφιλίωτα. Γι' αυτό ζητώ, κάνω έκκληση στην εισηγήτρια ώστε να ε, προσπαθήσει να μην ε, ξεφύγει από την πορεία της, από την πορεία που πρέπει να κρατήσει. Γιατί εδώ βάζουμε ε, στο κείμενο πράγματα που δεν πρέπει να μπουν. Έχουμε την αγορά. Η αγορά πρέπει να λειτουργήσει πρέπει να τις δώσουμε κάποια ελευθερία. Ε, και μετά το κομμάτι της υποχρεωτικής ταχυδρομικής ε, υπηρεσίας ε, έχει δημιουργηθεί για πολύ καλούς λόγους και καλό θα ήταν να μην πετάξουμε όλα τα καλά στοιχεία με μία ανάστροφη Λοιπόν, όσον αφορά το 4-1, εάν το βγάλουμε και δύο, εάν τα βγάλουμε τα στοιχεία αυτά, τότε δεν θα έχουμε ούτε και την καλύτερη ε, νομοθεσία, ούτε την καλύτερη ρύθμιση, δεν θα έχουμε τίποτα. Ε, ίσως ε, θα πρέπει να υποβληθούν άλλες τροπολογίες, γιατί η ποιότητα των συμβιβαστικών δεν είναι πολύ ψηλή. Κύριε Άντερσον, πρέπει ε, να τελειώνουμε. Ε, και εσείς ως εισηγήτρια, κύριε Άντερσον, έχετε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τη ρότα μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την έκθεσή της και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να βρει ε, κάποια κοινή γραμμή ανάμεσα από αυτές τις ε, διαφορετικές και αντιφατικές απόψεις. Γιατί είναι πολλές αντιφατικές απόψεις για το θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά για, τα, ε, για τις διεθνείς αποστολές είναι πολύ διαφορετική. Σε ορισμένες ε, αγορές, σε ορισμένες χώρες ε, η διαφάνεια είναι πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν όμως και άλλες χώρες όπου δεν ξέρουμε ακριβώς τι εφαρμόζεται. Ε, και δεν ξέρουμε και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες, ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς. Ε, πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη μεγαλύτερης ασφάλειας. Είτε μιλάμε για ιδιωτικές υπηρεσίες ή για δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή για υπηρεσίες εντός των δημοσίων υπηρεσιών ταχυδρομείου. Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι σαφής και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα η ρυθμιστική αρχή να παρεμβαίνει εάν και εφόσον υπάρχει στρέβλωση τη αγορά ή αθέμητο ανταγωνισμό. Ε, για να προστατεύσουμε κυρίως τις ε, μικρές μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει να δίνονται και εξάντε των προτέρων οι πληροφορίες ίσως στις εθνικές ρυθμιστικέ αρχές. Τώρα, όσον αφορά τι παρατυπίε. Και εδώ θα πρέπει να δίνεται στις εθνικές αρχές ε, αρκετή πληροφόρηση έτσι ώστε να αξιολογούν σωστά την αγορά. Υπάρχει ήδη το άρθρο 7 για το απόρριτο των στοιχείων και πιστεύω λοιπόν ότι μια και εδώ μιλάμε ε, για ε, ύπαρξη πολλών δεδομένων και στοιχείων, αυτό το άρθρο είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως ή πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφορές μεταξύ κρατών μελών ε, και φυσικά να έχουμε στόχο τη βελτίωση της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και βεβαίως να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτή την, την ε, περιπετειώδη ας πούμε πορεία της έκθεσης. Εδώ προσπαθούμε ε, να ε, συμφιλιώσουμε πράγματα ασυμβίβαστα. Από τη μία πλευρά έχουμε την υπηρεσία, την καθολική και υποχρεωτική υπηρεσία Ε, και τις δεσμεύσεις που έχουν αυτοί που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία και από την άλλη μεριά έχουμε την ε, εξέλιξη της αγοράς όπου αυτή η καθολική παροχή υπηρεσίας γίνεται όλο και λιγότερο αποδοτική. Ε, τα δέματα θεωρούν οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας ότι είναι τομέας προς ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά ε, ε, στην ουσία υπάρχει μια απειλή από πλευράς ε, των παρόχων καθολικής υπηρεσίας σε περίπτωση που θυγεί η αποδοτικότητά τους. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τη γενικότερη αποδοτικότητα της αγοράς και βλέπουμε ότι αν περάσουμε προς την ελεύθερη αγορά θα έχουμε προτάσεις οι οποίες θα ανταγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο, θα είναι αντίθετες προς τις ευαισθησίες του, της καθολικής ε, υπηρεσίας. Εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια αγορά η οποία απειλείται εντό εισαγωγικών ε, από τους, ε, από τους πάροχους σφαιρικών υπηρεσιών και εάν μιλήσουμε για αυτούς, τότε αν, απέναντί τους θα βρεθούν ενωμένοι και οι δημόσιοι πάροχοι και οι ιδιωτικοί ε, πάροχοι. Εν πάση περιπτώσει ε, βλέπουμε ότι οι απόψεις ε, δίστανται. Ε, τώρα δεν ξέρω ε, πώς μπορεί να γίνει η ψηφοφορία και τι αποτέλεσμα θα έχει, αλλά οπωσδήποτε θα αφήσει η κατάσταση αυτή μία πικρία, γιατί ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν ε, να διατηρηθεί ή ε, ο δημόσιος χαρακτήρας που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν πλήρως και έχουμε και αυτούς από την άλλη πλευρά που θέλουν να πάνε προς την ιδιωτική αντιμετώπιση που και αυτοί δεν μπορεί να ικανοποιηθούν πλήρως. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε, τουλάχιστον όχι μέσα από ένα τέτοιο εργαλείο, δεν θα καταφέρουμε να βρούμε έτσι μια κοινή συνιστόσα και η συγγήτρια παρά τις γενικές ε, παρατηρήσεις ε, κατανοούμε ότι ε, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη δυσκολία γιατί όλοι θέλουν την προστασία της καθολικής υπηρεσίας ενώ ταυτόχρονα θέλουν και ανταγωνιστικές τιμές ταυτόχρονα θέλουν και προστασία του καταναλωτή σε μια διευρυμένη και πιο απελευθερωμένη αγορά Τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω να, στην διαδικασία να κάνω εξειδικευμένε ε, παρατηρήσεις, να πω ότι θα πρέπει να ορίσουμε την ε, διαφάνεια ως εξή. Ε, οι ορισμοί άλλωστε για να ξεκινήσουμε δεν είναι ικανοποιητικοί. Νομίζω ότι εν τέλει ένα καλό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζήλερ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Άντερσον. Ε, δεν ήταν εύκολο το καθήκον της μέχρι τώρα. Όλα μια χαρά. Εγώ θέλω να μιλήσω για το 3 σχετικά με την ενημέρωση, του άρθρου 3. Κατά την άποψή μου, εδώ ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, πρέπει να, και μπορούμε να έχουμε κάτι που να ταιριάζει σε όλα. Υπάρχει το θέμα της ε, φορολογίας και πολλά παρεμπερί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω ως κατώτατο όριο να είναι οι 10 υπάλληλοι, η Λούση λέει 25. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι αυτό λύνει το πρόβλημα για όλα τα μικρά κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου θα θέλαμε η εθνική ρυθμιστική αρχή να επιλύει το θέμα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις ιδιαιτερότητες ε, των ε, κρατών ε, μελών. Να μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλου σε μόνιμη απασχόληση, μερική απασχόληση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να διευκολύνει τις εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν και το κοινωνικό dumping στη Λετωνία αν δεν πληρώνει κανείς τους φόρους, ε, έχουμε προβλήματα γιατί πολλές μεγάλες εταιρείες ε, αναθέτουν εξωτερική διεκπαιρέωση εργασιών ε, σε μικρές επιχειρήσεις. Εγώ όμως θεωρώ ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να έχουν κάποιες αρμοδιότητες να αποφασίζουν. Ο κύριος Μάρκος Φέμπερ που έφυγε μίλησε για τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις. Ε, να δούμε όμως ε, ποιες είναι αυτές που συμβάλλουν στην τεχνολογία. Στην Εστονία βλέπουμε μια εταιρεία η οποία σχεδόν χωρίς καθόλου υπαλλήλους, χωρίς καθόλου ηλεκτρονικά μηχανήματα να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Ε, μιλάμε για τέτοιου είδους νοφείς επιχειρήσεις και δεν είναι επικίνδυνο να υπάρχει κάποιο κατόφλι. Ε, πρόκειται για νεοφύς επιχειρήσεις με τεχνογνωσία, αλλά ε, βέβαια Ας πούμε στην Εστονία επιτρέπεται κάτι τέτοιο, σε κάποια πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμβαστική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Γκούλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ε, χαιρετίζουμε αυτό που ακούστηκε σήμερα, τη στήριξη στο άρθρο 3, δηλαδή την ε, βελτίωση του ρυθμιστικού ελέγχου, έτσι ώστε όλοι οι πάροχοι κάθε χρόνο να δίνουν πληροφορίες στις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Επίσης ε, χαιρετίζουμε το ότι προτείνονται κάποιες διευκρινήσεις όπως τον ορισμό του δέματος γιατί αυτό μεταξύ άλλων θα βοηθήσει στο να περιστεί το διοικητικό άκτος. Εξάλλου, συμφωνούμε και με αυτά που είπατε και εσείς σήμερα, ότι η αρχική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο άρθρο 4 δεν ήταν να επεκταθεί η διαφάνεια σε όλους τους παρόχους, αλλά μόνο οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών σε αυτούς να αφορά το άρθρο 4. Διότι με βάση αυτά που πιστεύει η Επιτροπή ε, θα πρέπει να υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη βάση που προβλέπεται στο άρθρο παριθμών 5. Ε, χαιρετίζουμε αυτά που ελέγχθησαν ότι είναι καλύτερα να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση Επιτροπής. Γιατί? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε άδικοι έναντι των παρόχων καθολικών υπηρεσιών αλλά για μας ε, το να υπάρχει εδώ δικαιοσύνη ε, σημαίνει ότι εστιάζουμε σε αυτούς, γιατί μόνο αυτοί έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες με προσιτό κόστος. Αυτό το σχέδιο κανονισμού ε, θεωρούμε ότι συμπληρώνει την οδηγία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών για να είμαστε σίγουροι ότι τα διασυνοριακά δέματα αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε το ότι υπάρχει σαφής αναφορά και στο άρθρο υπαριθμών 5 σχετικά με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 12 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Γιατί και πάλι για να μην υπάρχει μεγάλο βάρος στους, στις ρυθμιστικές αρχές έτσι ώστε και αυτές να εφαρμόζουν τις ίδιες αρχές όπως ισχύουν για την υπόλοιπη αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. Για να μην υπάρχει δεν πρόκειται για το στόχο. Νομίζω το περιεχόμενο του κανονισμού δεν αλλάζει το αντικείμενο των ε, καθολικών υπηρεσιών. Πράγματι, ε, ο στόχος ε, είναι ότι αυτό που θα έρθει μετά από δύο χρόνια να μην είναι αναθεώρηση, αλλά αυτό που θα έρθει μετά από δύο χρόνια θα είναι η έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών. Και, για τις, και τότε θα αναθεωρηθούν οι υποχρεώσεις των παρόχων καθολικών υπηρεσιών. Λυπούμεθα που διαγράφεται, προτείνεται να διαγραφεί το άρθρο 6, γιατί και πάλι Μπορεί να μην ήταν σαφή η αρχική διατύπωση, αλλά ο στόχο δεν ήταν να προβλέπεται υποχρέωση. Η υποχρέωση ήταν να γίνει κάτι. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να ε, απορρέει, να προκύπτει κόστος ε, για τους ε, λιανικούς εμπόρους, για τους λιανεμπόρους, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς, κύριε Άντερσον, ναι, έχω λίγα σχόλια. Ο Μάρκος Φέρντα έφυγε. Πάντως, να τον καθησυχάσω και πέστε αν τον δείτε, με κανένα τρόπο δεν ξεφεύγω από την καλή δουλειά που κάναμε για την οδηγία για τις αγιδρομικές υπηρεσίες και το σχετικό ψήφισμα ε, του περσινού χρόνου. Εμένω σε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά κάποια από αυτά, μέγα μέρος των θεμάτων που έχουν σχέση με την απασχόληση, χωρίς να τον ρυθμίζουμε, τον τομέα της απασχόλησης, πάντως έχει σχέση με στρεβλώσεις της αγοράς, όπως λέχθηκε και από άλλον. Θα επανέλθω σε αυτά, σχετικά με το τι κάναμε στις τελικές διατάξεις. Και βέβαια και η υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, συμφωνώ με τον Μάρκος Φέβερ ότι πρέπει και να προστατευτεί και να γίνουν σε αυτήν επενδύσεις. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έτσι ή δεν έρχεται σε σύγκρουση μαζί της. Κύριε Σλιτόφσκι, για την τροπολογία 282. Μπορούμε να επανέλθουμε και να δούμε στο κείμενο εάν υπάρχει τρόπος με τον οποίο θεωρείτε ότι τα συγκεκριμένα τιμολόγια μπορούν να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με την πρότασή σας. Αγνώσα το 282, μπορεί όμως να μην λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που προσπαθ, αυτόν προσπαθούμε να κάνουμε. Πάντως σας ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα σχόλιά σας. δεν πρόκειται για διπλασιασμό των δεδομένων, τα είπατε αυτά στα σχόλιά σας και έχετε δίκιο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε στο άρθρο 3 υποχρέωση που οδηγεί σε περιττή επικάλυψη δεδομένων. Και να συμφωνώ μαζί σας σε πολλά. Και πάλι δεν νομίζω ότι πάμε να φτιάξουμε κάποια νομοθετική ρύθμιση που να στρεβλώνει με οποιοδήποτε τρόπο την αγορά. Το λέω σε όλους και στον κύριο Ρικέ ότι θα πρέπει να μην δυσμονούμε ότι για τα δέματα στις περισσότερες χώρες μέλη αυτά έχουν μικρό μερίδιο της αγοράς των ε, ε, ε, επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται ήδη εκεί. Ψάχνουμε να βρούμε δεινόσαυρους δηλαδή, αν, ψάχνουμε, αν προσπαθούμε να βάλουμε τη ρύθμιση μόνο σε αυτό το θέμα, χωρίς να περιλάβουμε όσο γίνεται περισσότερα σχετικά με τους νέους επιχειρηματίες. Και δεν θέλω να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε Συμφωνώ με αυτά που λέτε ότι είναι πολύ φιλόδοξη η προσπάθεια αυτή. Αλλά επειδή είναι συγκεκριμένο θέμα, μόνο διαμεθοριακού χαρακτήρα και μόνο για δέματα, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Και για εσά, Βιμ, δεν προσπαθώ να συμβιλώσω τα συμφιλίωτα, ελπίζω ότι είναι δυνατόν να συμφιλειωθούν και θα εξακολουθήσει να παραμένει απλό και λιτό. Ε, δεν προτείνω άλλα δέκα άρθρα, πραγματικά όχι. Θα μείνει λοιπόν απλό και λιτό και υποστηρίζω και την αρχή της βελτιωμένης νομοθεσίας. Κάθε τι που πράττουμε λοιπόν θα το ελέγξουμε και θα, θα το διπλοελέγξουμε για να είμαστε βέβαιες ότι είναι σωστό. Για την Κλάουδια, σωστό αυτό που είπατε, πρόκειται για ζητήματα δικαιοσύνης, φέρνες και για την ενή αγορά και πώς να διαμορφωθεί αυτή σωστά. Είπατε επίσης ότι οι ρυθμιστικές αρχές ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους από άλλες. Βρισκόμαστε εδώ πράγματι στην Ευρώπη, σε μια κατάσταση ευρωπαϊκή. Και η οδηγία για τι εκδρομικέ υπηρεσίε δεν έχει δημιουργήσει πλαίσιο που να επιτρέπει σε όλε τι ρυθμιστικέ αρχέ να πράττουν ό,τι πρέπει. Ορισμένε ναι, ορισμένε όχι. Αυτό είναι μια περιορισμένη πτυχή του θέματο. Ουδή ισχυρίζεται ότι θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά όλα δια Για το άρθρο 3, ας εξετάσουμε τις παραπέρα προτάσεις σας, πώς μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε τη διακριτική ευχέρεια στις χώρες μέλη για ορισμένα ζητήματα του απασχολούμενου προσωπικού. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σχόλια. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που ε, φαίνεται όλους τους απασχολεί το θέμα και όλοι το προσέχουν. Σας ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 11η Ιουλίου. Πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε καλές συμβιβαστικέ λύσεις και έτσι ώστε να ακουστεί ο λόγος του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε προχωρήσει γρήγορα. Euh, θα σας προτείνω ένα διάλειμμα, γιατί το άτομο με το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε δεν έχει έρθει ακόμα. Πέντε λεπτά διάλειμμα λοιπόν.

Λοιπόν, οδική ασφάλεια. Ασφάλεια οδικών μεταφορών δηλαδή. Έχουμε εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση MOVE σχετικά με την εφαρμογή οδικών τεχνικών ελέγχων βάσει του κανονισμού 0116 και 0099. Ε, μιλάμε για την περίοδο μέχρι το 14 και θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία. Θα σας πω αμέσως σε ποιον θα δώσω το λόγο. Okay. Είναι εκπρόσωπο της Επιτροπής, σας το πούμε έτσι πιο γενικά. Είναι η κυρία Ιωαννίδου. Ιωαννίδου. Κοιτάξτε, λέει η κυρία Ιωαννίδου, θα σας ε, παρουσιάσω μία γενική άποψη του ε, εγγράφου, το οποίο αφορά τους οδικούς ε, ελέγχους για τα εμπορικά οχήματα από το 13 μέχρι το 14 αυτή είναι η περίοδος βεβαίως ε, στην Eurlex υπάρχει διαθέσιμη η πλήρης έκθεση, το πλήρες κείμενο δηλαδή ε, κάθε δύο χρόνια ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των ελέγχων που έχουν κάνει, τα γνωρίζετε αυτά και πρέπει να πω ότι τούτη τη φορά τα κράτη-μέλη είχαν κάποιες ε, ε, αργοπορίες. Υπήρχαν βέβαια και μερικές χώρες ε, οι οποίες ε, υπέβαλαν έγκαιρα. Έχουμε με κίτρινο τις αργοπορημένες και κάποιες χώρες οι οποίες δεν συμμορφούνται. Διότι, και σας εξηγώ γιατί. Διότι τροποποιήθηκε η οδηγία του 2000 με μία του 2010 βάσει της οποίας προβλέπονται κάποιες νέες διαδικασίες αναφοράς και αυτή ήταν η πρώτη αναφορά που έγινε ε, με τις ε, νέες ε, προδιαγραφές ας πούμε. Υπήρξαν δυσκολίες για κάποιες χώρες, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά και είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη έκθεση θα είναι πλήρως συμμορφωμένη. Εδώ βλέπετε ποια είναι η κατανομή των ελέγχων μεταξύ ιδιωτικής χρήσεως και μη ιδιωτικής χρήσεως, δημοσίας χρήσεως, καθώς επίσης και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες ε, χώρες βλέπετε ότι τα στοιχεία είναι ε, διαφοροποιημένα. Άλλε φορέ έχουμε την ε, επεξήγηση, άλλες φορές λείπει η επεξήγηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ε, βάσει αυτής της περίοδου ε, και βάσει των αριθμών των ελέγχων είπαμε ότι, είδαμε ότι οι έλεγχοι μειώθηκαν κατά 31% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το συζητήσαμε αυτό με την Επιτροπή Ελέγχου των, των ε, δρόμων ε, ε, το προηγούμενο Μάιο και αυτοί μας έδωσαν διάφορες εξηγήσεις. Πρώτον, μας είπαν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου είχαν άλλες προτεραιότητες και το, η δεύτερη εξήγηση είναι λίγο καλύτερη, ότι δηλαδή ορισμένες φορές η μείωση του αριθμού των ελέγχων ε, οφείλεται σε καλύτερες ε, ε, μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί και πιο στοχευμένες μεθόδους. Αυτό είναι θετικό και αποτελεί θετική εξέλιξη, εξέλιξη διότι σημαίνει ότι δεν χάνουμε χρόνο με ανώφελους ελέγχους θα μπορούσα να αναφερθώ και σε συγκεκριμένες χώρες, αν θέλετε μπορώ να το κάνω αργότερα. Τώρα, σε αυτό το γράφημα βλέπετε ε, τους αριθμού, τον αριθμό απαγορεύσεων ε, ε, οχήματα των οποίων απαγορεύτηκε η κυκλοφορία μετά τους ελέγχους. Ο αριθμός αυτών των οχημάτων έχει αυξηθεί. Το 2011-2012 είχαμε 5,1 ενώ τώρα έχουμε 9,8 Βλέπετε πάντως ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα που για μία ακόμα φορά μας οδηγεί ε, στο ερώτημα κατά πόσο είναι αποτελεσματική η στοχευμένη έλεγχη και αν η στόχευση είναι σωστή. Επίσης, ε, σε γενικές γραμμές τα ιδιωτικά οχήματα φαίνεται να ε, μάλλον ε, τα οχήματα τα οποία έχουν αγοραστεί και κυκλοφορούν ε, στην ημεδαπή συντηρούνται καλύτερα από αυτά που έχουν αγοραστεί και συντηρούνται στην ελλαδαπή. Εδώ βλέπετε τα, τα κυριότερα προβλήματα και αναποτελεσματικότητες που αναφέρουν τα κράτη-μέλη. Εδώ εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Μπορεί, υπάρχουν τα στοιχεία Πάντως σημειώνουμε ότι ορισμένες ε, χώρες ε, παρουσιάζουν ε, περισσότερο κάποια συγκεκριμένα ελαττώματα ή ελλείψεις. Περνάω τώρα στην επόμενη διαφάνεια σας παρακαλώ. Τα συμπεράσματα λοιπόν. Αυτά είναι τα κύρια, τα τρία κύρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συγκρατήσετε από τούτη την έκθεση. Πρώτον, μείωση του αριθμού των ελέγχων επιθεωρήσεων, ε, μείωση κατά 31,5%, το ανέφερα ήδη και προηγουμένως. Εάν συστηματικά ε, είχαμε μαζί με τη μείωση αυτή και ε, αυτόματα αύξηση των ε, οχημάτων τα οποία έχουν, για τα οποία έχει απεκορυφθεί η κυκλοφορία, αυτό θα ήταν θετικό και είναι. Τώρα η ισορροπία, αυτό είναι το τρίτο στοιχείο, ανάμεσα στα ημεδαπά και αλλοδαπά οχήματα, αλλά η ισορροπία δεν είναι σωστή πάντα σε όλα τα κράτη-μέλη, σε ορισμένες χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά ε, σε άλλες περιπτώσεις η κατάσταση πόρο απέχει από το να είναι ικανοποιητική. Τέλος, έχουμε το ζήτημα της αναλογίας ε, των απαγορευμένων οχημάτων είναι πολύ μικρή, ε, μικρό ποσοστό του 0,5%, πράγμα που σημαίνει ότι η στόχευση δεν είναι αποτελεσματική και επομένως χάνουν οι εταιρείες πολύτιμο χρόνο. Και επίσης αυτό καταδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριμένες χώρες ε, ε, πολύ ψηλά ποσοστά, 89% για ε, μεταγράφα οχήματα σε μια συγκεκριμένη χώρα. Το θέμα της στόχευσης λοιπόν, καλύτερη στόχευση, αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα οδηγία που θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη χρονιά και η οποία εισάγει ένα καλύτερο σύστημα αξιολόγησης κινδύνου και επομένως ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια θα οδηγηθούμε σε καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερη εναρμόνιση. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. κύριε Ιωαννίδου. Για να δούμε ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. Βιμ Βαντενκάμπ. Ε, ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Μην ε, εκλάβετε εσφαλμένα αυτό που θα πω, αλλά θα πρέπει να διαβάσω την παρουσίαση αυτή μαζί με την ε, δέσμη μέτρων περικινητικότητας για να την κατανοήσω. προτείνεται αύξηση των ελέγχων στους δρόμους κατά 3% όλων των δράσεων. Δεν είναι βέβαιο αν αυτά 3% θα στοχεύουν την αποκάλυψη του καμποτάζ ή θα είναι τεχνικού χαρακτήρα. Πρώτη ερώτηση λοιπόν αυτή. Δεύτερη. Ποια είναι η κατάσταση της ενσωμάτωσης της εθνικές υπηρεσίες επιθεωρήσεων. Υπάρχει μια εθελοντική συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών επιθεωρήσεων, η e ΑΣΥ νομίζω λέγεται, European Route Control δηλαδή. Πώς λειτουργεί η συνεργασία αυτή μεταξύ των επιθεωρητών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτο, είναι απογοητευτικό που δύο, οι μη δύο μείζονες χώρες μέλη, η Γερμανία και η Γαλλία, ε, δεν κατόρθωσαν ή δεν θέλουν να ανακοινώνουν, βέβαια δεν είναι ερώτηση, το σημειώνω απλώ δεν κάνουν report. Τώρα έχω και μια πιο ολλανδική ερώτηση. Έχει κάπως λαϊκό χαρακτήρα, λαϊκίστικο χαρακτήρα θα έλεγα μάλλον, αλλά στις κάτω χώρε υπάρχει εντύπωση ότι η έλεγχη είναι αυστηρότερη για εύπορους Ολλανδούς οδηγών φορτηγών από ότι για λιγότερο εύπορους και φτωχούς οδηγούς φορτηγών από άλλες χώρες. Έχει κάτι να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και Βάντεν Κάμπ. Εσείς κυρία μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελαμβάνω το λόγο επειδή υπήρξα εισηγήτρια εδώ στο Ευρωκοινοβουλίο για την οδηγία, για τη συγκεκριμένη οδηγία και ομολογώ ότι η σημερινή παρουσίαση θυμίζει πολύ τη συζήτηση που είχαμε διεξαγάγει προετών και τότε είχαν πει έλεγχοι και επιθεωρήσεις πρέπει να είναι πιο στοχευμένοι γιατί καμιά φορά υπάρχουν υποψίες διακριτικής μεταχείρισης και μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών μελών. Άρα αυτά δεν είναι νέα στοιχεία, ούτε προκαλούν καμιά έκπληξη. Αυτό που ήθελα να πω ήδη λέχθηκε από τον ε, κύριο Βάντε Κάμπ. Στην ουσία την ίδια ερώτηση θα ήθελα να θέσω. Οι χώρες μέλη από τις οποίες χρειαζόμαστε τα αριθμητικά δεδομένα, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, γιατί δεν τα δίνουν. Τι κάνουμε με αυτό. Δεύτερη ερώτηση σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου. Και αυτό ακριβώς θέλαμε, για το λόγο αυτό ακριβώς θέλαμε να περιληφθεί. Θέλουμε στοχευμένες επιθεωρήσεις, στοχευμένες ε, επί των πιο επικίνδυνων μεταφορέων. Και το 2019 θα γίνει εισαγωγή του συστήματος. Οι χώρες μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν να αρχίσουν να λειτουργεί δηλαδή το σύστημα ε, από το 2019. Αυτό νομίζω πρέπει να επιδιώξουμε. Ε, εσείς κύριε ε, Ολλανδικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ έχω ερωτήσεις παρόμοιας κατευθύνσεως. Η έλεγχη. Έχει κάνει κάποια ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει την περίοδο αναφοράς. Την περίοδο των αναφορών δηλαδή. Και οι χώρες μέρη θέλουν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για να είναι πιο αποτελεσματική. Τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητέ. Είναι πολύ ενισχυτικό που οι δύο μεγάλες χώρες δεν είναι σε θέση να υποβάλουν εκθέσεις. Θα το δεχθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα αναλάβει δράση. ώστε να υποβάλλονται στο μέλλον εκθέσεις. Διότι η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων έχουν θεσπιστεί στην νομοθεσία. Υπάρχουν, ε, προβλέπονται οι υποχρεώσεις αυτές. Θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον πρόκειται για συστηματική διαδικασία, να μπορεί να προσφύγει, να κινήσει διαδικασίες για παραβίαση. Κύριε Κράμερ, εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την έκθεση. Για την παρουσίαση δηλαδή που είναι κάπως απογοητευτική. Χαίρομαι που μάθαμε τώρα ότι η Γερμανία και η Γαλλία ουδόλως ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται κάτι να γίνει. Εσείς στο κάτω της γραφής είστε οι θεματοφύλακες των συνθήκων και της οδηγίας. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορείτε απλώς να λέτε, α, ναι, εντάξει, δεν μας δίνουν τα δεδομένα, ωραία και μετά θα ξανακούσουμε έκκληση και θα μάθουμε πάλι ότι δεν δίνουν τα δεδομένα οι δύο αυτές χώρες. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεύτερο, τα όσα εξετάζονται, συμφωνεί, βρίσκουν να λείπει κάτι. Το 10% των φορτηγών είναι παραφορτωμένα. Έχετε στατιστικές για αυτά τα πράγματα. Είναι πάλι η Γερμανία και η Γαλλία οι δύο χώρε που δεν δίνουν τα σχετικά δεδομένα. Κάνατε κάποια προσπάθεια, υπάρχουν πίνακες. Θα ήθελα να το γνωρίζω. Διότι τα υπερφορτωμένα φορτηγά είναι μεγάλος κίνδυνος. Και για τους ίδιους αλλά και για όλους τους υπολείπους. Τρίτο, ε, ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης. Είχαμε πάει σε ένα σταθμό ελέγχου και εκεί μας είπε η αστυνομία Χτες ένας οδηγός μας είπε παρακαλώ ελέγξτε με 17 ώρες είμαι στο τιμόνι και ο, το αφεντικό δεν μου επιτρέπει να κάνω ε, ε, διάλειμμα. Και ξέρουμε ότι αυτά συμβαίνουν συχνά. Άρα εφαρμογή του νόμου χωρίς ελέγχους, ξεχάστε το. Το ερώτημα είναι τι γίνεται εκεί και εκεί ε, πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ε, ελέγχους σε ποσοστό 0,1%. Τι γίνεται, τελευταίο βλέμμα στο μέλλον. Μιλήσαμε για το ντίζελ. Και αν έχουμε τώρα για τους φόρους επί του diesel, real driving emissions, τι θα γίνει εκεί ή και αυτά είναι ε, στα μάτια. Αλλά γνωρίζουμε τι έχουν κάνει οι μηχανικοί για να καταστατηγήσουν τις νομοθετικές προβλέψεις. Αυτό είναι το όραμα για το μέλλον. Τι θα κάνει πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς το βλέπετε. Γιατί και αυτό είναι μέγας κίνδυνος. Ευχαριστώ αγαπητέ Κράμερ. Βλέπετε ότι οι ερωτήσεις θέτουν το δάκτυλο επί των τύπων των είδων. Δεν λέμε και ποτέ, θα το, ποτέ ότι ένας νεκρός στους δρόμους, ένας θάνατος στους δρόμους, σημαίνει άλλα 7 πρόσωπα τα οποία μένουν ανάπηρα. Βαρύτατο κόστος για ε, την κοινωνία. Αυτή η υπόθεση των μεταφορέων, των οδικών μεταφορών. Νομίζω εδώ το πραγματικό ζήτημα, το είπαν και όλοι άλλωστε, είναι το ζήτημα των ελέγχων. Εγώ ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει η κυρία Τελή, εκ παραδρομής. Ως πρόεδρος της Επιτροπής, εννοώ βεβαίως. Ακόμα δεν έχω γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάντως, δηλώνω συγκλονισμένη. Όπως είπε ο κύριος Βαντεκάμπ, στην δέσμη μέτρων για την κινητικότητα δεν είναι τίποτα για τον έλεγχο αλλά θα περιμένουν λέει το 2034. 2034 και μέχρι τότε πρώτο σχόλιο. Δεύτερο και λέχθηκε από τον κύριο Κράμερ ο έλεγχος του χρόνου αναπαύσεως αλλά και των συνθήκων αναπαύσεως των οδηγών όταν έχετε μεταφορείς που κοιμούνται μέσα στις καμπίνες των φορτηγών σε συνθήκες πραγματικά αφόρητες. Ε, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις σήμερα στο 2017. Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, διότι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξεκουραστεί είναι επικίνδυνος. Και επικίνδυνο να προκαλέσει βαρύτατα ατυχήματα. Τέλος, διαφάνεια. και το μέγα διακύβημα για την Επιτροπή μας, ώστε οι μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, ακόμα δεν έχουν υποβάλει εκθέσεις, ακόμα δεν έχουν διαθέσει τα δεδομένα τους για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε τα ερωτήματα αυτά, αν μπορείτε λοιπόν, θαύμα θα είναι, κυρία Ιωαννίδου, Ιωαννίδου, θα είναι θαυμάσιο. Και μετά θα δώσουμε και το λόγο στον κύριο Λιεζουά. Ε, πιο εύκολα το λέω αυτό, Λιεζουά. Ορίστε, Λοιπόν, ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα των δύο μεγάλων ε, κρατών μελών για να είμαστε απόλυτα σαφείς. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι αυτά τα κράτη-μέλη δεν μας έδωσαν στοιχεία. Ε, πιστέψτε με, την κάνουμε τη δουλειά μας, την κάνουμε καλά. Μας έδωσαν στοιχεία, αλλά δεν είχαν τα στοιχεία ολοκληρωμένα, γιατί υπήρχαν και κάποιες ε, νέες ε, ταξινομήσεις με βάση την ε, τροπολογία υπαρτιμών 10. Ήταν αναγκασμένα τα κράτη να τροποποιήσουν τα, τις, τα δεδομένα ή τον τρόπο που συλλέγουν τα δεδομένα και μας είπαν ότι θα μας ενημερώσουν με βάση τους νέους κανόνες. Το θέμα είναι ότι έχουμε γενικά τα δεδομένα, αλλά μας λείπουν κάποιες κατηγορίες δεδομένων. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής ότι και τα δύο κράτη συνεργάστηκαν, γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, να μην κάνουμε την τρίχα τριχιά ε, και εμείς ε, κάναμε τη δουλειά μας και εκείνοι έκαναν τη δική τους. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι συζητάμε για τις τεχνικές επιθεωρήσεις. Εστιάζουμε την προσοχή μας στα ελαττώματα και τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα οχήματα. Υπάρχει εδώ κάποια σύγχυση, γιατί υπάρχουν άλλες επιθεωρήσεις που αφορούν στο ωράριο εργασίας και αυτό το θέμα θα σας το παρουσιάσει ο συνάδελφός μου ο Έντι, ο οποίος είναι αρμόδιος για το δέσμι μέτρων για την κινητικότητα. Ως εκ τούτου αυτό που αναφέρατε για το 3% δεν ισχύει εδώ. Ε, σας λέω, εμείς μιλάμε για τα τεχνικά προβλήματα των οχημάτων, μόνο γι' αυτό. Κατά τα ε, δεν ε, έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μας ε, για διακριτική μεταχείριση, αυτό δηλαδή που έθιξε ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής. Και συμφωνούμε τα με την κυρία Σενχάνοβα και ζητώ συγγνώμη αν δεν προέφερα καλά το όνομά σας. Είναι αλήθεια ότι η αξιολόγηση κινδύνου είναι ένα θέμα κλειδί, είναι οδηγία εξετάζει το θέμα αυτό και με βάση την επόμενη έκθεση θα ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη να προβούν σε πιο στοχευμένες επιθεωρήσεις. Ε, την πρώτη συζήτηση την κάναμε ήδη το Μάιο και δεν ξέρουμε τώρα να σας πούμε κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα ε, προχωρήσουν πιο γρήγορους ελέγχους, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα ασκήσουμε πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά στο θέμα των παραφορτωμένων ε, φορτηγών. Ε, πρέπει να σας πω, λυπάμαι πολύ, αλλά αυτό είναι εκτός ε, της κείμενης νομοθεσίας, γιατί η νομοθεσία εξετάζει, λέω, μόνο τα τεχνικά προβλήματα. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω στοιχεία. Ναι, αλλά αυτό που σας είπα εγώ είναι πιο σημαντικό από τα τεχνικά προβλήματα. Δυστυχώ δεν έχω στοιχεία από αυτού. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ ο συναδελφό σας. Θα απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις και μετά θα περάσω στην ε, παρουσίαση του επόμε... της επόμενης έκθεσης. Να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα λοιπόν όσον αφορά την επιβολή του νόμου είναι ένα σημαντικό σημείο προς ε, βελτίωση ε, στην ε, δέσμη κινητικότητας. Το αντιμετωπίσαμε αυτό, δέσμη της 31ης Μαρτίου. Ε, και ε, επίσης ε, και στον άλλο κανονισμό για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδηγού μεταφορέα. Επίσης θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό κυρίως λόγω της ύπαρξης των πλασματικών ψευδεπίγραφων ας πούμε εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, λέμε ότι θα πρέπει να ε, ζητούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από κάθε εταιρεία και να, κάνουν, γίνονται και επιτόπιοι έλεγχοι. Ο κύριος Βαντενκάπ αναφέρθηκε στο ποσοστό ελέγχων που θα πρέπει να διεξάγονται στο μέλλον ανακράτος μέλος. Αυτό το ποσοστό ε, εάν ε, θυμάμαι καλά αυτό το 6% σχετίζεται με το καμποτάζ μόνο. Ε, εμείς ε, προτείνουμε να αλλάξει ο κανόνας του καμποτάζ, να απλουστευτεί και το κατόφλι όριου του καμποτάζ, αλλά πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται και κάποιοι ελάχιστοι έλεγχοι ε, καμποτάζ. Ε, και με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί και ο ίδιος ο κανόνας, αλλά ε, από την άλλη πλευρά το κράτος μέλος θα αναλάβει την ευθύνη να κάνει ε, ελάχιστο αριθμό ελέγχων που έχει οριστεί στο 3% για το καμποτάζ στο έτος μείον 2. Επίσης, να σας πω ότι οι πληροφορίες που θα, δώσουν, που θα καταχωρήσουν τα κράτη-μέλη στο ε, Μητρό, ιδίω δε ο, το, ο αριθμός ε, πεδίου καταχώρησης ε, ε, του φορτηγού και της οδικής μεταφοράς θα λαμβάνονται υπόψη γιατί ξέρετε ότι υπάρχει διασύνδεση και επομένως έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις οδικές μεταφορές. Αυτά είναι ορισμένα από τα μέτρα τα οποία εμείς προτείνουμε. Κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε Επίσης, ε, στην ανάπαυση εντός ε, του ε, φορτηγού αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό στο κείμενο, στην νομοθεσία για την οδήγηση και την ανάπαυση. Εμείς προτείνουμε να μειωθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπαυση μπορεί να λάβει χώρα εντός του φορτηγού και ε, λέμε ότι επί των ωρών εργασίας 45 ώρες τουλάχιστον θα πρέπει ε, να, ε, να είναι ο οδηγός εκτός του φορτηγού και με τον τρόπο αυτό να μπορεί κάθε τρεις εβδομάδες τουλάχιστον να γυρίσει και στο σπίτι του. Όσον αφορά τους ταχυγράφους, Ε, και όσον αφορά και την, ε, ε, την, το, την νομοθεσία 2034 του 2017 όσον αφορά τους ευφυείς ταχυγράφους τώρα για την ώρα ασχολούμαστε με την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού και θα ακολουθήσουν οι τεχνικές ε, ε, εξειδικεύσεις για τους ε, ταχυγράφους και μετά και για, ταχυγράφους και μετά για τους ευφυείς ταχυγράφους Μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερον, όπως είπατε και εσείς, δεν υπάρχει υποχρέωση retrofit Όσοι καταγραφούν πριν από τον ε, Ιούνιο του 2017 ε, θα μπορούν να προχωρήσουν στον ψηφιακό ταχογράφο που δεν είναι ακριβώς ο εφής αλλά είναι μια εξέλιξη. Ε, να σας πω επίσης ότι έχουμε ξεκινήσει μία έκθεση, μία έρευνα μάλλον, μελέτη, όπου θα μελετήσουμε τις ε, διαφορετικές ε, ε, περιπτώσεις εφαρμογής retrofit πριν πριν υπάρξει γενικευμένη χρήση των εφιών των Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό απήντησα στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε κάτι σε σχέση με την ερώτηση του κυρίου Βαντανκάμπ σχετικά με αυτό το 3%. Είπατε ότι υπάρχει τροποποίηση του καμποτάζ, αλλά ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο ε, ποσοστό καμποτάζ. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποια είναι η τροποποίηση σχετικά με το καμποτάζ. Τι εννοείτε όταν λέτε τροποποίηση καμποτάζ. Γιατί δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Θα ήθελα λοιπόν να μου το πείτε αυτό. Τι εννοείτε συγκεκριμένα όταν λέτε τροποποίηση του καμποτάζου, κύριε Βαντενκάμπ. Κύριε... Κυρία Πρόεδρε, για να καταλάβω κι εγώ και να ξέρουμε και για το μέλλον, έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα καλά όταν γίνεται επιθεώρηση ενός φορτηγού, τεχνική ε, επιθεώρηση και κοινωνική επιθεώρηση γίνονται ταυτόχρονα. Είναι σωστό ή δεν κατάλαβα καλά. Άλλες ερωτήσεις. Monsieur Liégeois, vous avez deux questions. Έχετε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα να απαντήσετε. Έχετε τη δικιά μου και την ερώτηση του κύριου Βαντανκάμπα. Θα ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του κύριου Λιεζουά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκα σε μια τροποποίηση του κανονισμού ε, του ορίου για το καμποτάζ. Ε, μέχρι τώρα ε, οι μεταφορείς μπορούν να κάνουν τρεις συναλλαγές καμποτάζ τρεις μέρες μετά μια διεθνή μεταφορά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο τριών συναλλαγών καμποτάζ και επομένως υπάρχει ένας περιορισμός που σύμφωνα με την πρότασή μας εκφράζεται μονάχα με χρονικούς όρους. Ένας λοιπόν ε, εμπορευόμενος μπορεί να κάνει συναλλαγή καμποτάζ στις πέντε μέρες, πέντε μέρες μετά, ε, την, μετά από μια διεθνή συναλλαγή στο κράτος μέλος. Euh, επομένως, επομένως, αφαιρέσαμε το, τον περιορισμό ε, σε σχέση με τον αριθμό των ε, συναλλαγών ε, και γιατί είδαμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν οδηγούμαστε σε απελευθέρωση του καμποτάζ. Εμείς, σύμφωνα με την πρότασή μας, μειώνουμε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας μπορεί να λάβει χώρα το καμποτάζ. Από τις 7 πάμε στις 5 μέρες. Και για να σας ξαναεξηγήσω, το μέτρο ελέγχου ε, είναι ε, απολύτως καινούριο, δεν υπάρχει στην υφιστάμενη ε, οδηγία. Τα κράτη-μέλη σύμφωνα με, την, με τον νέο κανόνα λοιπόν πρέπει, οφείλουν να κάνουν ένα τουλάχιστον 3% ελέγχους στις συναλλαγές καμποτάζ και ως περίοδο αναφοράς ε, παίρνουμε το έτος μείον 2 έτσι ώστε ε, να ορίσουμε τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων καμποτάζ. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές κάνουν ελέγχους που καλύπτουν διάφορα νομοθετικά ζητήματα, ας πούμε και διάφορα κείμενα, ας πούμε ε, ε, σεβασμός του όσον αφορά τον ταχογράφο και όσον αφορά την κοινωνική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικέ ήθελε να υποβάλει ένα ερώτημα, κάτι που δεν κατάλαβα καλά ε, για το καμποτάζ. Πριν είχαμε μια διάρκεια χρονική επταήμερη. Είχα, υπήρχε λοιπόν το δικαίωμα αυτό επί σειρά 7 ημερών. ήταν 7 εργάσιμες μέρες ή 7 ημέρες ε, μετρώντας τη μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια της ε, ε, εργάσιμης ή μη ημέρας. Ας πούμε ότι είναι ημερολογιακές ημέρες, τις παίρνουμε τη μία μετά την άλλη. εργασιμης η ημερας ας πουμε οτι μέρες ήταν για το καμποτάζο στο κράτος μέλος. Ο κύριος Ρικέ. Ε, οι αδειοδοτήσεις κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων δεν έχουν όμως απαγόρευση κυκλοφορίας αυτών των βαρέων οχημάτων δύο μέρες τη βδομάδα εκτός από ειδικά ευαίσθητα εμπορεύματα. Κοιτάξτε, ο μεταφορέας οφείλει να σεβαστεί τις, ε, ε, τους περιορισμούς κυκλοφορίας που νομοθετεί το κράθε, κράτος μέλος. Εάν σε αυτές τις 7 ημέρες, μία ή περισσότερες μέρες, σύμφωνα με το κράτος μέλος στο οποίο κυκλοφορεί, ε, υφίσταται απαγόρευση κυκλοφορίας, πρέπει να τη σεβαστεί. Δεν μπορεί να κάνει ούτε διεθνή συνδιαλλαγή, ούτε συναλλαγή, ούτε μπορεί να κάνει και συναλλαγή καμποτάζ. Ναι, κοιτάξτε, αλλά αυτή η απαγόρευση κυκλοφορία ε, στο Σαββατοκύριακο ε, ισχύει για όλε τι χώρε μέλη. Επομένω, ε, σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να υπάρχει καμία συναλλαγή. Επομένω, ήδη μιλάμε για 7 μέρε και από τι 7 περνάμε στι 5. οι 5 αυτέ οι μέρε. σημαίνει ότι ε, έχετε απελευθέρωση του καμποτάζ. Γιατί από τις 7 μέρες από τις οποίες τις 2 δεν μπορούσαν να γίνουν συναλλαγές, περνάτε στις 5 ελεύθερες ημέρες. Το πέρασμα λοιπόν από 7 σε 5 μέρες, λαμβάνοντα υπόψη ε, την απαγόρευση κυκλοφορίας ε, των δύο ημερών ανά εβδομάδα, σημαίνουν ότι δεν άλλαξε καθόλου η κατάσταση και δεν, άλλαξε, δεν μειώθηκε καθόλου το καμποτάζ αλλά ανταποκρίνεται στην ε, θέση που είχε πάντα η Κομισιόν, δηλαδή της πλήρους απελευθέρωσης του καμποτάζου. Ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Είναι το τελευταίο μας σημείο. Αφορά παρουσίαση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενός κατεξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνω τον λόγο στην κυρία Ιζαμπέλ Βαντών η οποία είναι επικεφαλής της ε, μονάδας ε, καινοτόμων μεταφορών. Έχετε τον λόγο κυρία μου. Bonjour. Euh, peut-être pourrais-je d'abord parler la... επιτρέπετε να δώσω πρώτα το μικρόφωνο στον διευθυντή μου, ο οποίος έχει κάνει τη μετακίνηση και μετά να προχωρήσω. Πώ τον λένε το διευθυντή σα που όλοι τον γνωρίζετε, αλλά εμείς όχι. Τράιτος ή κάπω έτσι. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς Ισαμπέλ που με επιτρέπετε να λάβω πρώτο το λόγο. Για να πω κυρία Πρόεδρε ότι πρόκειται ένα εγχείρημα σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι για να προσαρμοστεί η κατεξουζότηση πράξης έχει γίνει συνάντηση με τους εμπειρογνώμες του Κοινοβουλίου στα πλαίσια της οδηγίας ITS για έκτη φορά νομίζω τώρα με κατεξουζότηση πράξη επαναλαμβάνω που πραγματικά η κυρία Βαντών θα σας παρουσιάσει με πλήρη γνώση μιας και είναι η αρμοδία θεματάρχης του αφήνω λοιπόν, ε, της επιτρέπω μάλλον, αν επιτρέπετε εσεί να λάβει το λόγο για να σα εξηγήσει την κατεξοχή πράξη που πολύ σύντομα θα εφαρμοστεί. Να μου επιτρέψετε να συνεχίσω τα αγγλικά γιατί ξέρω καλύτερα την ορολογία. Πρόκειται για την εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίθηκε μέσα στη δέσμη μέτρων κινητικότητα 31 Μαΐου και τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο εξετάσεω, scrutiny period. Όπως είπε ο διευθυντή μου, ο έχουμε διάφορες δράσεις προβλέψει για να διασφαλίσουμε συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και των χωρών μελών και του Κοινοβουλίου που είχαν προσκληθεί σε μια νέα ομάδα εργασίας για να συντάξουν το κείμενο μέσα σε 11 συνεδρίες ανάμεσα στο Νοέμβριο του Μαρτίου και στον ε, Μάιο ε, ναι, το, Μάρτιο του 2016 και είχαμε και δύο εβδομάδες επιγραμμικής διαβουλεύσεως μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2015 είχαμε και μια υποστηρικτική μελέτη Αυτά έδειξαν θετική επίπτωση. Κάναμε και πολλές διμερείς επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, του stakeholders δηλαδή, για να εξασφαλίσουμε ότι η την πράξη θα είναι ικανοποιητική για όλους. Μιλούμε εδώ για πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων για ταξίδια με στόχο ταξιδιωτικούς σχεδιασμούς μέσα από όλους τους τρόπους μεταφορών. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω access points εθνικών. Θα μπορούν να διοχετεύονται τα δεδομένα αυτά κατά φάσεις και να υπάρχει ελευθερία και το καθήκον να εγκρίνουμε ποιοι θα, ποιοι θα είναι οι μορφές που θα λαμβάνουν τα εθνικά access points. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι τα δεδομένα θα πρέπει να είναι τυποποιημένα στα εθνικά access point. Ο κατεξουσιώτης κανονισμός περιλαμβάνει εναρμονισμένο σύνολο μορφοτύπων μέσα από τους διάφορους τρόπους μεταφορών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ε, μεταφραστικά σετ για να μπορέσουν να περάσουν αυτά στις διάφορες ε, γλώσσες. Ένα άλλο θέμα που ήταν σημαντικό στις συζητήσεις μας ήταν οι όροι και προϋποθέσεις για τις άδειε, καθώς και ποιοτικά κριτήρια που συναποτελούν μέρος του κατεξουδότησης κανονισμού. Όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς operator μεταφορών. Τα δεδομένα θα παρέχονται για το σύνολο των μεταφορικών δικτύων, πληροφορίες όπως χρονοδιαγράμματα, ε, τρόποι πρόσβασης, προσβασιμότητα για πρόσωπα με μειωμένη ικανότητα και ούτω καθεξής θα πρέπει να έχουν δοθεί μέχρι το 2019 πληροφορίες για bike sharing, για δηλαδή κοινή χρήση των αυτοκινήτων και ούτω καθεξής θα πρέπει να έχουν ε, δοθεί μέχρι το 2020 πιο λεπτομερείς πληροφορίες για παράδειγμα για ποδηλατικά δίκτυα, για ε, κατεκτήμηση ε, ώρες αφήξεως κλπ. μέχρι το 2021 για το συνολικό δίκτυο μέχρι το 2023. Αυτά είναι τα ε, ε, στατικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τα δυναμικά δεδομένα, δηλαδή πραγματική, πραγματική χρόνη μάλλον πού βρίσκεται τώρα ο σύρμος μου, το τρένο μου και ούτω καθεξής. Μετά από τις διαβουλεύσεις κατέληξαν οι χώρες μέρη ότι θα τα κρατήσουν αυτά στα, σε δική τους αρμοδιότητα, στα εθνικά access point και αν το πράξουν αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Η κατεξουσιώτηση πράξη επιτρέπει πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά όχι μόνο. Επιτρέπει και τον σχεδιασμό ταξιδιών μέσω διασύνδεσης υπηρεσιών στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όταν υπάρχει ζήτηση. Δεν υποχρώνουμε λοιπόν όλες τις Travel Information Services να διασυνδέονται, όμως όπου υπάρχει ζήτηση υπάρχει υποχρέωση απάντηση στη ζήτηση. Συνιστούμε επίσης την χρήση ευρωπαϊκών interface, των EPI, καθορίζουμε ε, τα σημεία όπου θα μπορεί να ψάξει κανείς να βρει πού αρχίζει το ταξίδι, πού τελειώνει, πού πρέπει να γίνει η διασύνδεση, καθώς και συμβατικές ε, ε, συμφωνίες. Σε βάση συμβάσεων δηλαδή. Για να τα κάνουμε αυτά έχουμε προγράμματα στήριξης της διευκόλυνσης δηλαδή, στην Ευρώπη ως μέρος του προγράμματος εργασιών του 2016. Έχουμε ξεκινήσει τώρα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τις χώρες μέλη με άμεσες επιχορηγήσεις και 100% συγχρηματοδότηση για τις χώρες μέλη με 5 εκατομμύρια που θα μοιραστούν οι χώρες μέλη για να καλύψουν διάφορες διαστάσεις της κατεξουσιοδότησης πράξης. Οι δε χώρες μέλη μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με την κατάστασή τους αν θέλουν να επενδύσουν σε stakeholder engagement, σε εκπαίδευση, σε διασπορά των πληροφοριών. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να φτιάξουν τα access point ή για να τα διευρύνουν, αυτά που υπάρχουν ήδη για παράδειγμα για τα δεδομένα των οδικών μεταφορών ή για την οδική ασφάλεια. Αν θέλουν να χρηματοδοτήσουν διαλειτουργικότητα, δηλαδή να μετασχηματίσουν τοπικά δεδομένα στους μορφοτύπους που προβλέπονται για τα δεδομένα ή αν θέλουν να προωθήσουν τον συνδυασμένο σχεδιασμό ταξιδιών. Αυτά μέχρι τέλος του έτου. Και μετά μπορούν να αρχίσουν οι χώρε μέλη την εργασία από τον Ιανουάριο του 2018. Η ιδέα δραστηριότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Αυτό ολοκληρώνει την ε, παρουσίασή μου. Έχουμε και άλλε διαφάνειε, εάν θέλετε, με περισσότερε λεπτομέρειε αλλά αν θέλετε μπορούμε να διακόψουμε εδώ και να κάνουμε συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση σας. Έχετε ερωτήσεις εσείς οι ευρωβουλευτέ. Κύριε Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω ότι καταρχήν εγώ δεν είμαι ειδικό για αυτά τα θέματα. Ίσως τώρα οι ερωτήσει μου να μην είναι οι απόλυτα ενδεδειγμένες, αλλά το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει κατεξουσιοδότηση κανονισμός. Ξέρω ότι είναι κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά κατεξουσιοδότηση κανονισμός αυτό δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Από πού έρχονται τα δεδομένα. Ποιος δίνει δεδομένα σε ποιον. Από τους ε, φορείς ε, παροχής ε, σιδηροδρομικών υπηρεσιών, από ποιους. Και το τρίτο μου ερώτημα, ποιος ωφελείται από όλα αυτά. Ο μεμονωμένος ε, καταναλωτής αναφέρθηκε η διαλειτουργικότητα, η πολυτροπικότητα. Μπορείτε λιγάκι να μου εξηγήσετε γιατί εδώ ε, αυτά έχουν σχέση και με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Μπορείτε να μου τα εξηγήσετε και ποιο βοηθάει ποιον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εντάξει, ούτε κι εγώ είμαι ειδικό, όπως είπε και ο κύριος ε, και ο προλαλής σας, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και ε, νομίζω ότι Σαφής ήταν η εισήγηση. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι τα ε, στατικά δεδομένα, το χρονοδιάγραμμα, όπως επίσης και το δυναμικό χρονοδιάγραμμα. Και διερωτώ με πώς φτάσαμε τελικά στα δεδομένα ε, το 2020, το 2021 ε, σε σχέση με τη μελέτη του 2019. Άλλη μία προβλέπεται για το 2021 αν θυμάμαι καλά, και έχει σχέση με τους ε, ποδηλατόδρομους με τον εκτιμόμενο χρόνο ταξιδιού. Υπάρχει ένας λόγος γιατί προτείνεται αυτό το χρονοδιάγραμμα. Το 2020 και το 2021 θα τηρηθούν ή ε, θα μπορούσαμε να πάμε και λίγο πιο νωρίς. Το δεύτερο είναι κάτι που με απασχολεί. Το πρόγραμμα δράσης 5 εκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν σε 27-28 κράτη-μέλη. Μπορώ να φανταστώ ότι θα έχουμε ένα δάνειο της τάξης το 100% αν αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, διότι μπορούμε να πιστεύουμε ότι το κράτος μέλος ε, είναι διστακτικό και θέλουμε να προχωρήσει το όλο εγχείρημα. Είναι ένα είδος κινήτρου. Έχετε 4-5 στόχους και ο καθένας μπορεί να επιλέξει. Στην πραγματικότητα λοιπόν Αν δεν υπάρχει συνέργεια, κατανοώ ότι η Κομισιόν μπορεί να πει ότι αυτά είναι καθοριστικά και θέλουμε αυτά να είναι ο στόχος, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι μετά από πέντε χρόνια θα υπάρχει κάποια δυσαναλογία. Υπερβάλλω, αλλά θα υπάρχει κάποια δυσαναλογία σχετικά με το κόστος, το εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ για 4-5 στόχους μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές. Κατανοώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, 150 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ίσως κάτι να μην κατανοώ στο στόχο. Και πρέπει να σας πω ότι νιώθω κάπως άβολα αν κάποιος μας ρωτήσει γιατί ε, καταρτίζεται αυτός ο προεπλογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας λέω, ίσως να μην κατανοώ κάτι, αλλά ψάχνω να δω την αποτελεσματικότητα. Κατά τα άλλα, θα δούμε πώς όλα αυτά μπορούμε να τα συνδέσουμε με το να είμαστε πιο κινητική μέσα από την ε, πολυτροπικότητα. Ελπίζω να ήμουν και εγώ εξίσου αδαή στο θέμα αυτό, όσο και ο κύριος Βαντεκάμπ. Ο κύριος Κράμερ. Σας ευχαριστώ για την ε, εισήγησή σας, αλλά έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, το θέμα των ε, integrated ticketing. Αυτό το αποφασίσαμε πριν από 10 χρόνια στη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Είπαμε ότι ε, μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, αλλά μετά από 10 χρόνια η πραγματικότητα είναι ότι αυτό δεν ισχύει. Στα αεροπλάνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσε αεροπορικέ εισιτηρίε και αν εμπλέκονται δεν ε, έχω πρόβλημα. Όμω όχι στου σιδηροδρόμους. Και αυτό το ε, θεωρώ ένα εγωιστικό λάθος. Γιατί οι εταιρείε σιδηροδρόμων ε, λένε όχι εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τα στοιχεία μας αλλά με τον τρόπο αυτό βλάπτουν και τους άλλους. Πρέπει λοιπόν να σκεφτεί πίεση. Εγώ θέλω να έχω ε, πληροφορίες σε ολόκληρο τον κόσμο αν θέλω να ταξιδέψω με τους, με το σιδηρόδρομο, όπως γίνεται και με το αεροπλάνο εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με τα αεροπλάνα, δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματικό πόρτο, γιατί να υπάρχει και για τους ε, σιδηρόδρομους. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγχρηματοδοτούνται. Και ερωτώ, ε, μπορούμε να έχουμε πληροφορίες ε, σχετικά με τα προγράμματα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα προγράμματα είναι ολοκληρωμένα ή όχι. Γιατί αν έχουμε τρεις-τέσσερις ε, διαφορετικές έρευνες ε, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Μετά, όσον αφορά την πώληση των εισιτηρίων, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, πολύ ενδιαφέρον, τι γίνεται με το διοξίδιο του άνθρακα από τις Βρυξέλλες έως τη Μαδρίτη. Αν πάρω το αεροπλάνο γνωρίζω. Αυτές είναι οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Αν πάρω το αυτοκίνητο επίσης, αν πάρω το, το ποδήλατο και το πλοίο τα γνωρίζω ή πρέπει να τα γνωρίζω και ο πελάτης να ξέρει ότι το καθοριστικό θέμα δεν είναι μόνο η τιμή αλλά και η διάσωση του περιβάλλοντος. Και ρωτώ γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Και επειδή ήδη χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, Εν τω μεταξύ συμβαίνει το εξή στου σιδηρόδρομου, αν πρόκειται και μπλέκονται δύο χώρε, μπορώ να κλείσω online ένα εισιτήριο. Αν όμω είναι τρει οι χώρες, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή από τις Βρυξέλλες παίρνω το Ταλής στο, στο Παρίσι, από το Παρίσι το βραδινό τρένο για τη Μαντρίτη. αυτό όμως δεν μπορώ να το αγοράσω σε ένα εισιτήριο ε, γιατί είναι τρεις οι χώρες και δεν το καταλαβαίνω, αλλά αυτό που σας λέω αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ακόμα πιο τρελή είναι η κατάσταση. Εγώ ξέρετε ότι είμαι τρελός με το ποδήλατο. Και αν πάω από το Βερολίνο προς το Άμστερνταμ με Intercity, μπορώ να το κλείσω online. Αν πω όμως ότι θέλω από το Βερολίνο προς το Άμστερνταμ να πάρω το ποδήλατό μου παρότι στο Intercity μπορώ να πάρω το ποδήλατο, δεν μπορώ να κλείσω ηλεκτρονικά για το ποδήλατο. Τρελό και αυτό, δεν ξέρω γιατί, αλλά και αυτό είναι διακριτική μεταχείριση των τουριστών που χρησιμοποιούν ποδήλατο. Και γιατί γίνεται αυτό. Νομίζω λοιπόν αυτή είναι δουλειά της Κομισιόν ίσα δικαιώματα για όλους. Ε, Παραδείγματος χάρη, ε, με τα αυτοκίνητα. Μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου από το Βερολίνο προς τη Βιέννη ή τη Ζηρίχη, αλλά και παλαιότερα, ακόμα και πριν από 20 χρόνια, ε, κάναμε διαδήλωση γιατί σε αυτά τα ε, τρένα μπορεί να βάλει κανείς το αυτοκίνητο, τη μηχανή, αλλά όταν εγώ ήθελα το ποδήλατο, μου είπαν όχι, ποδήλατο απαγορεύεται. Γελάει ο κύριος από την Κομισιόν και αυτός είναι φανατικός του ποδηλάτου, αλλά εγώ σας λέω, για ε, δικαιώματα για όλους, ό,τι ισχύει για τα χοντροαυτοκίνητα δεν μπορεί να μην ισχύει για τα ποδήλατα και τώρα περιμένω με μεγάλη αγωνία την απάντηση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Στρέφομαι προς την ε, Κομισιόν κύριε Αντέρση. Ευχαριστώ. Βεβαίω, ε, λέω στον κύριο Βαντεκάπ ε, ότι μπορούν να υπάρξουν ε, κατά εξουσιοδότηση πράξης μετά τη θέση ισχύ. Γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση πως έχει. Για τα άλλα σχόλια σχετικά την χρήση αυτού του φακέλου των 5 ε, εκατομμυρίων είναι συγκεκριμένη και στοχευμένη η στόχευση. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν έχουν προχωρήσει όλα ε, στον ίδιο βαθμό. Σε άλλα έχουν ήδη δημιουργηθεί οι δομές, σε άλλα ε, όχι. Υπάρχουν πολλές στοχευμένες δράσεις οι οποίες ε, θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το grant του 100%. Ε, το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να διασπαρούν τα χρήματα αυτά στις 27 χώρες σε μικρό ε, πράγματα. Ε, όσον αφορά τώρα την το επιγραμμικό κλείσιμο εισιτηρίων, καθώς επίσης και το κατά πόσο μπορεί κανείς να πάρει το, αερο, συγγνώμη, ποδήλατό του, ε, να πω το εξή ε, ε, η Ιζαμπέλ γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, ίσως πρέπει εκείνη να απαντήσει. Να επανέλθουμε στο πιο δίνει τι. Όλοι οι μεταφορείς, είτε είναι δημόσια αρχή, είτε και ένα ιδιωτικό car sharing, ε, μπορούν να δώσουν τα ε, στοιχεία. Εάν εγώ μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, των στοιχείων που πρέπει να ε, να, δίνονται. Σας βεβαιώθηκε ότι θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει απόρριτο, δεν ζητούμε κάποιες πληροφορίες ας πούμε. Ε, αλλά πιο πολύ, σε ποιο σταθμό πήρατε ε, το κόσμο, ε, πόσο κοστίζει, ποιος είναι, ποιο είναι το εκτιμόμενο μέσο κόμιστρο, τέτοιου είδους ερωτήσεις. Και εφαρμόζονται επίσης και στις αεροπορικές μεταφορές, στο μετρό, στον προαστιακό, στα ε, πλοία λοιπά. Ε, και στα λεωφορεία ακόμα. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία? Όλοι. Διότι θα γίνουν open data. Βεβαίως ε, θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες όμως απλώς θα κάνουν λόγο στο είδος χρήσης ε, μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα, μπορεί να είναι επιχειρήσεις, ε, οποιοδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα την έχει. Όσον αφορά ε, το τίμημα, στη δημόσια διαβούλευση το συζητήσαμε αυτό Ε, αποφασίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα planning το οποίο να είναι καλό και αντιμετωπίσιμο ας πούμε από όλους. Τίποτα παραπάνω από αυτό. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε όσο γίνεται ε, περισσότερο με συνένεση. Τη συνένεση προσπαθούμε να βρούμε. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι το planning, ε, ε, ο σχεδιασμός για ταξίδια που περνάνε από πολλές ε, χώρες είναι όντως κάτι πιο περίπλοκο. Εμάς, εμείς δουλεύουμε με κόμβους. Θα ξεκινήσουμε με το συνολικό δίκτυο Comprehensive Network και θα βλέπετε λοιπόν εκεί όλες τις μεγάλες πόλεις που καλύπτονται από το δίκτυο σχετικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μπορούν, μπορεί να δοθεί το ισοδύναμο των εκπομπών, αλλά ακόμα ε, δεν είναι υποχρεωτική αυτή η αναφορά στον κανονισμό. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα στοιχεία. Monsieur Reuters, Madame je vous Σας ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία ε, σας εδώ και την παρουσίασή σας και βεβαίως είστε πάντα καλοδεχούμενοι εάν θελήσετε να ξαναέρθετε. Ο κύριος Κράμερ θέλει να ρωτήσει κάτι. Έχω μια ερώτηση ακόμα. Είχαμε μιλήσει παλαιότερα για το πακέτο Αλτεμαν. Εάν οι συνδρομικές επιχείρησεις δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν εντός τριετίας ότι θα έχουμε όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη, τότε θα το πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ το είχα βρει καλή ρυθμίση αυτή διότι είχαμε σκεφτεί θα αντιδρούν, θα αντιδράσουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Θα κάνουν κάτι ή θα κάνουν τίποτα και τότε θα δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικώς τι έγινε. Εσείς κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως κύριε Κράμερ. Μόλις τώρα μπήκε το πακέτο σε εφαρμογή και μέχρι το 2019 έχουμε χρόνο να δούμε αν οι stakeholders θα αντιδράσουν. Η κατεξουσιοδότηση στην πράξη αποτελεί κατάλληλο συμπλήρωμα. Αναμένουμε λοιπόν πολλές δράσεις που θα ξεκινήσουν από αυτήν την κατεξουσιοδότηση στην πράξη. Θα παρακολουθούμε επί μία τριετία πολύ προσεκτικά και θα δράσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Βάουτερς. Έχετε άλλες ερωτήσεις εσείς οι ευρωβουλευτέ. Κύριε Τέλινσκα, μία μικρή ερώτηση. Σύντομη δηλαδή. Πολύ σύντομα. Περισσότερο μια συνέχεια μετά από αυτό που είπε ο κύριος Κράμερ. Κατανοώ πλήρως ότι δεν αποτελεί στόχο της κατεξουσία της συμπράξεως αλλά με την ευκαιρία απευθύνομαι στον διευθυντή που γνωρίζω ότι και γνωρίζει αλλά έχει και προοδευτικό πνεύμα, να στο πω έτσι, για το integrated ticketing. Φτάνουμε σιγά σιγά ε, στο τέλος της κοινοβουλευτική μας εντολής, αλλά εκτός από την ε, έκθεση πρωτοβουλίας δεν έχουμε άλλες προσπάθειες. Κάτι θα χρειαστεί να γίνει. Όλοι μας περιμένουμε ότι θα έχουμε το integrated ticketing σε λίγα χρόνια, δύο-τρία χρόνια. Αυτό που αναμένουμε όμως είναι να ξεκινήσει η διαδικασία και αυτή να είναι σταδιακή. Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα σημεία εχμής στην ε, προσπάθεια για το ολοκληρωμένο εισιτήριο. Αναμένω λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδυάσουν τις προσπάθειές των και να γίνει τουλάχιστον ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το ονειρευόμαστε και μιλούμε γι' αυτό χωρίς να έχουμε καμιά ορατή εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι λοιπόν ακριβώς ερώτηση, αλλά δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το θέμα του integrate και την επειδή δεν μπαίνει στην κατεξουδότηση στην πράξη. Δεν εντάσσεται δηλαδή. Ευχαριστώ εσείς κύριε Ρόιτερς. Θα είμαι σύντομος κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ όμως με ε, την φιλοξία του κύριου Βουλευτού. Όντως χρειάζεται ανάρρευση δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα είπε άλλωστε στο Mobility Package, ότι θα ε, το εντάξει στα δικαιώματα των επιβατών και των ε, επιβατών πολυτροπικών μέσων και την κινητικότητα ως υπηρεσία που τα βάζουμε, τα εντάσσουμε στην ψηφιακή αυτή εξέλιξη. Και γνωρίζω ότι αυτά ενδιαφέρουν πολύ την Επιτροπή σας καθώς και την πρόεδρό Έχουμε και συνάντηση ε, τέλη Δεκεμβρίου στο Ταλίν και η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί για τις πολυτροπικές μεταφορές με τη σαφή φιλοδοξία να κάνουμε περισσότερα για το αντικείμενο αυτό που ούτε εύκολο είναι και είναι και περισσότερο, ε, εντάσσεται περισσότερο στις υπηρεσίες αλλά έχει μια σαφή φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή που τονίσατε και εσείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτερς. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα κηρύξω το τέλος της συνεδριάσεως και ήταν όντως το τελευταίο θέμα αυτό. Κύριε Βαντεκάμπ, μην είστε θλιμμένος, θα ξαναειδωθούμε στις 10 Ιουλίου. Μην ανησυχείτε. Από τις 10 και μετά. Θα είστε παρόν. Και εσείς και εμείς.